So, uh, dear colleagues, ladies and gentlemen, it's already a few minutes past so I propose to start our meeting of today. Κυρίες και κύριοι, προτείνω να ξεκινήσουμε, έχουν περάσει κάποια λεφτά, οπότε προτείνω να ξεκινήσουμε. Καθίστε παρακαλώ, για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, πρώτο θέμα, έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, εγκρίνεται. Δεν βλέπω να υπάρχουν αντιρρήσεις, ενστάσεις. Δεύτερο θυμία, έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων της 23 η και 24 η Ιανουαρίου 2017. Αν δεν υπάρξουν σχόλια μέχρι το τέλος της σημερινής μας συνεδρίασης θα θεωρηθούν ότι εγκρίνονται. Τρία. Ανακοινώσει του Προέδρου σχετικά με τις αποφάσεις που έλαβαν οι συντονιστές. Αποφάσεις που ελήφθησαν από τους συντονιστές στη συνεδρίαση τους της 23ης ε, Ιανουαρίου έχουν συμπεριληφθεί στα πρακτικά της σχετικής ε, συνεδρίασης. Θα θεωρηθούν εγκεκριμένα εκτός αν υποβληθούν ενστάσεις στη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης. 4. Ανακοινώσει του Προέδρου Έχω διάφορε ανακοινώσει να κάνω σήμερα. Πρώτον, ως συνήθως, η συνεδρίασή μας μεταδίδεται στο διαδίκτυο και έχουμε διερμηνία. Για τη διευκόλυνση των διερμηνέων, Σα παρακαλώ να μιλάτε αργά. Έχω και μια ανακοίνωση που αφορά έναν ε, συνάδελφο, τον κύριο Γκάουκλας Κογέλτη δυστυχώς εγκαταλείπει τη γραμματεία της ε, Επιτροπής ΙΝΤΑ έπειτα από 5,5 χρόνια λόγω απαιτήσεων κινητικότητας προσωπικού και θα ήθελα εκ μέρους των μελών της ε, Επιτροπής ΙΝΤΑ να του ευχηθούμε κάθε επιτυχία στην, ε, στα νέα του καθήκοντα στην γραμματεία της Επιτροπής ΑΦΕΤ. Και φυσικά είναι πάντοτε καλό να γνωρίζουμε ότι υπάρχει κάποιος πρώην συνάδελφός μας στην Επιτροπή αυτή, στην ΑΦΕΤ, ο οποίος θα γνωρίζει καλά τα δικά μας θέματα. Υπάρχουν και διάφορα ε, νέα που αφορούν το εμπόριο της ε, προηγούμενης περίοδου. Πρώτον, η Συμφωνία Διευκόλυνση Εμπορίου που τέθηκε σε ισχύ. Πρόσφατα εγκρίθηκε η συμφωνία αυτή από, το, από τη Ρουάντα, το ΟΜΑΝ, το Τσάντ και άλλες χώρες. Υπάρχουν πλέον πάνω από 110 χώρες του ΠΟΕ που έχουν εγκρίνει αυτή τη συμφωνία. Αυτό σημαίνει ότι το όριο που απαιτούνταν για να τεθεί σε εφαρμογή η ε, συνθήκη, η συμφωνία αυτή έχει επιτευχθεί τρία χρόνια μετά την ε, σύνοδο του Μπαλί. Η συμφωνία αυτή θα ενισχύσει τη διαφάνεια, τον ε, προσδιορισμό προδιαγραφών, την μείωση των τελών, ιδίως για τις αναπτυσσόμενες χώρες. Και υπάρχουν εκτιμήσεις ότι θα υπάρξει έως και 15% μειώσεις για τις εμπορικές συναλλαγές στις φτωχότερες χώρες. Η συμφωνία αυτή έχει και πολιτική σημασία διότι καταδεικνύει την σημαντικότητα ε, της ε, πολυμερούς συνεργασίας και ε, της αμοιβαίας ωφέλειας στις παγκόσμιες εμπορικές συναλλαγές. Το Κοινοβούλιο ενέκρινε την προσχώρηση της Ένωσης το Σεπτέμβριο του 2015. Ο, ο, εξέδωσε πρόσφατα ε, κατευθυντήρες γραμμές για τα ενδύματα και τα υποδήματα και την ε, λειτουργία των, της αλυσίδας τροφοδοσίας για την ε, εξασφάλιση της ε, δέουσας επιμέλειας. Έχουν υπάρξει συνεισφορές και συμβολές τόσο από τις επιχειρήσεις όσο και από τους εργαζόμενους και από τις οργανώσεις κοινωνίας των πολιτών και έτσι καταρτίστηκαν οι κατευθυντήριες γραφές, γραμμές αυτές και έχουμε και μια σχετική γνωμοδότηση για την ε, Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για τον τομέα των ενδυμάτων που θα συζητήσουμε. Συμφωνία Τρίψη για την βελτίωση της πρόσβασης ε, σε φάρμακα τέθηκε σε εφαρμογή την 31η Ιανουαρίου. Δύο τρίτα των μελών του ΠΟΕ έχουν πλέον ε, εγκρίνει αυτήν την τροπολογία στη συμφωνία αυτή, αναγνωρίζοντας ότι τα μέλη του ΠΟΕ θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν προβλήματα τα μέλη εκείνα τα οποία δεν έχουν ή έχουν πολύ ε, χαμηλή συνεισφορά στον, ε, κλάδο των φαρμάκων. τα περισσότερα φάρμακα που παράγονται ε, με ε, εγχώρια άδεια μπορούν να διατίθενται μόνο στις αγορές των χωρών στις οποίες παράγονται. Αυτό ε, δυσκολεύει την διάδοση των γενώσιμων φαρμάκων, κάτι που είναι απαραίτητο για την αντιμετώπιση των προβλημάτων δημόσιας υγείας που αντιμετωπίζουν οι φτωχότερες κυρίως χώρες. Αυτή η τροπολογία στην Συμφωνία TRIPS του ΠΟΕ ε, είναι η πρώτη σημαντική αλλαγή ε, από το 1995 οπότε και συμφωνήθηκε το συγκεκριμένο κείμενο. Και τελευταίο νέο, ε, υπάρχουν διαπραγματεύσεις εμπορικού χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με δύο χώρες της Ασίας, την Ινδονησία και τις Φιλιππίνες. Ο δεύτερος γύρος των συζητήσεων με την Ινδονησία ξεκίνησε στα μέσα του 2016 ε, και συνεχίστηκε τον Ιανουάριο του 2017. Η Ινδονησία είναι η μεγαλύτερη αγορά της Νοτιοανατολικής Ασίας με ε, περισσότερο από 250 εκατομμύρια κατοίκους και συνεχίζονται οι συζητήσεις για το SPS, το DBT, την διακίνηση αγαθών, τις ε, κρατικές προμήθειες, την βιώσιμη ανάπτυξη, την επίλυση διαφορών και άλλα θέματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δημοσιεύσει τις 9 διαπραγματευτικές της προτέσεις. Αυτές παρουσιάστηκαν και στις ε, Φιλιππίνες κατά το δεύτερο γύρο συζητήσεων που έγινε πριν από δύο εβδομάδες. Οι Φιλιππίνες είναι η δεύτερη μεγαλύτερη χώρα της ε, περιοχής με πληθυσμό άνω των 100 εκατομμυρίων ανθρώπων. Επόμενο θέμα της σημερινής διάταξής μας είναι η κατάσταση των συνεχιζόμενων διαπραγματεύσεων του τριμερούς διαλόγου. Όσον αφορά τις ε, συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις έχω τη χαρά να σας πω ότι οι διοργανικές διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο και την Κομισιόν θα ξεκινήσουν σχετικά με το εργαλείο ε, για, την, ε, για την εμπορική άμυνα με τον εισηγητή μας. Οι συζητήσεις ε, είναι υπερόριμες καθώς η πρόταση της Κομισιόν είχε υποβληθεί τον Απρίλιο του 2013 και το Κοινοβούλιο ενέκρινε τις τροπολογίες της την επόμενη χρονιά το Φεβρουάριο του 2014. Λόγω της, ε, των εργασιών ε, του, στο Συμβούλιο είχαμε μάλιστα ολοκληρώσει την πρώτη ανάγνωση της πρότασης πριν την λήξη της προηγούμενης ε, του Κοινοβουλίου. Τώρα, πλέον μπαίνουμε στο δεύτερο ε, γύρο συζητήσεων με σκοπό να ολοκληρωθούν οι συζητήσει το συντομότερο δυνατό. Η συγκητή μα δεν είναι εδώ σήμερα. Δεν ξέρω αν υπάρχουν σχόλια που θα ήθελε να υποβάλει κάποιο σε σχέση με αυτό το θέμα. Δεν βλέπω. Επομένως, περνάω αμέσως στο σημείο 6 που είναι η αξιολόγηση των εξωτερικών παραμέτρων της τηλεονιακή επίδοση και διαχείρισης ω μέσο διευκόλυνση του εμπορίου και της καταπολέμησης του λαθρεμπορίου. Η συγγήτριά μα είναι η κυρία Τιτσιάνα Μπεγκίν και με έχουν ενημερώσει ότι η έκθεση της εισηγήτριας ε, έχει λάβει 126 τροπολογίες για τη βελτίωσή της. Ωστόσο πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι ε, θα πρέπει να έχουμε στο επίκεντρο της προσοχής μας μόνο τα ζητήματα που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες της Επιτροπής μας. τροπολογίες βρίσκονται στο στάδιο της εξέτησης και κάποιες ενδέχεται μάλιστα να μην εμπίπτουν στο πεδίο των αρμοδιοτήτων μας. Γι' αυτό και ο Πρόεδρος ε, εξετάζει το ενδεχόμενο να ε, χαρακτηρίσει ορισμένες από τις τροπολογίες που έχουν υποβληθεί ως απαράδεκτες. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στην Τιτσιάνα για να μας παρουσιάσει την έκθεσή της. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συναδέλφοι, καταρχάς θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για το ενδιαφέρον που δείξατε για το θέμα αυτό και μάλιστα ε, αυτό αποδεικνύεται και από τις 126 τροπολογίες που ανέφερε προηγουμένως ο Πρόεδρος. Αυτό αποτελεί παράδειγμα του ενδιαφέροντος που υπάρχει για το θέμα αυτό. Επομένως χαίρομαι παρά το γεγονός ότι κάποιες μπορεί να μην ε, ε, γίνουν δεκτές. Εγώ θεωρώ ότι πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό θέμα διότι η καλή λειτουργία των τελωνίων μας ε, αποτελεί πυλώνα της κοινή εμπορικής πολιτικής. Η ομοιόμορφη λειτουργία τους ε, είναι ικανή και αναγκαία συνθήκη ώστε να έχουμε πραγματικά μια εμπορική πολιτική όπως ε, πολύ σωστά είπαμε και είναι γνωστό της πάση. Ε, είναι κατακαιρματισμένες οι ευρωπαϊκές πολιτικές και αυτό δημιουργεί προφαινόμενα τα οποία είναι εις βάρος των πολιτών μας και των επιχειρήσεών μας, κυρίως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ε, της παραγωγής στην Ευρώπη, η οποία κινδυνεύει από την παραποίηση και το παράνομο εμπόριο. Όσον αφορά την προθεσμία για την κατάθεση των τροπολογιών, έκανα μία σειρά από επισκέψεις ε, σε ευρωπαϊκά και ιταλικά λιμάνια για να έχω μια πιο ε, ε, συγκεκριμένη εικόνα του πώς έχει κατάσταση, να συναντήσω και τους εργαζομένους του τομέα και να δω και όλους τους ενδιαφερομένους. Και Διαπίστωσα, όπως είχα και στο παρελθόν, ότι υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ των ευρωπαϊκών λιμένων ώστε να προσελκύουν εμπορεύματα από τρίτες χώρες. Και αυτό όχι μόνο ε, με βάση ε, τον θεμητό ανταγωνισμό, αλλά επωφελούμενοι και κάποια κενά στην νομοθεσία. Επομένως, ε, έχει δύο όψεις το φαινόμενο. Υπάρχουν εισαγωγείς και εξαγωγείς οι οποίοι προτιμούν ένα λιμάνι γιατί υπάρχουν λιγότεροι έλεγχοι και λιμένες οι οποίοι ανταγωνίζονται στις παρυφές της νομιμότητας για να μπορέσουν να ευνοήσουν τελικά αυτές τις συμπεριφορές. Χαίρομαι λοιπόν που διαπιστώνω ότι και η τροπολογία σας έχουν αντίστοιχες ανησυχίες, όπως Επίση, διαπίστωσε και ότι υπάρχει ευαισθησία για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και την απλούστευση του γραφειοκρατικού άχθου. Στην πραγματικότητα από τις 126 τροπολογίες ελάχιστες ε, με βρίσκουν αντίθετη. Θα προσέξω όμως πάρα πολύ, θα τις συζητήσω στις επόμενες συνεδριάσεις και θα δούμε από εκεί και πέρα εάν ε, θα γίνουν παραδεκτές ή όχι. Ε, πολλές άλλες τροπολογίες όμως με βρίσκουν απόλυτα σύμφωνοι να υπενθυμίσω κάποια θέματα τα οποία είναι πολύ σημαντικά κατά την άποψή μου. Το γεγονό ότι πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένε πληροφορίε για τον τύπο των ελέγχων που διεξάγονται στα τελωνία, όπως επεσήμαναν οι σοσιαλιστές και οι δημοκράτες, την ανάγκη να εναρμονίσουμε ε, τους τύπους των ελέγχων, ε, τροπολογίες που υπέβαλε ε, η ομάδα των φιλολευθέρων. ο ιδιωτικό τομέα ο, ο οποίος... Ε, απασχόλησε το ECR. Επίσης πρέπει να υπάρχει μηχανοργάνωση και να είναι διαλειτουργικά τα συστήματα ελέγχου και να μπορέσουμε να έχουμε και κατάλληλους πόρους για να υλοποιηθούν αυτά. Αυτό το ανέφεραν και το ΕΛΚ και οι σοσιαλδημοκράτες, καθώς επίσης και ανάγκη να γίνει αξιολόγηση των εμπορικών ροών ε, λόγω μιας ε, ε, επιλογής ενός λιμένα ο οποίος μπορεί να είναι πιο βολικός αλλά μπορεί να είναι πιο ε, ε μακριά από γεωγραφικής άποψης όπως επεσήμενε οι πράσινη. Υπάρχουν και κάποιες τροπολογίες που με βρίσκουν πάρα πολύ σύμφωνοι. Την ανάγκη να δούμε ότι η διαδικασία για τη δέουσα επιμέλεια γίνεται σεβαστή. Συνάδελφοι, πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να βλύνουμε τις διαφορές μας και θα μπορέσουμε να υποβάλουμε μία πρόταση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την επίλυση του προβλήματος αυτού που με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο πλήττει τους συναδέλφους. Ε, είμαι στη διάθεσή σας λοιπόν για να ακούσω σχόλια και παρατηρήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Και τώρα να δώσουμε το λόγο στους κοιόδης ηγητές, εξ του ΕΛΚ, ο κύριος Μπένσιν. Καταρχάς, ε, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω. Δεν έχω πολλά επί της από πλευράς του ΕΛΚ. Απλούστευση και μείωση του γραφειοκρατικού άχθους ε, είναι πάρα πολύ σημαντικά για μας, αλλά νομίζω ότι αυτά καλύφθηκαν και σε προηγούμενες συζητήσεις. Επομένως, ε, θα είμαι πάρα πολύ σύντομος. Ε, προσβλέπουμε στο πρώτο σχέδιο συμβιβαστικών τροπολογιών από την εισηγήτρια και από ό,τι κατάλαβα από τα όσα μας είπε σήμερα μπορεί να δεχτεί τις περισσότερες από τις τροπολογίες. Ε, περιμένουμε λοιπόν τις τροπολογίες και ίσως θα μπορούσε η εισηγήτρια να μας πει και πότε θα μπορούσαμε να περιμένουμε και μια πρόταση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Για τους σοσιαλιστές και δημοκράτες, ο κύριος Σούστερ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ε, αντικαθιστώ την ε, αρμόδια σχεδόν του μας, την κυρία Οντρίγκες Ριμπέρο, και να σας πω λοιπόν τα εξή εξ, της, ότι, εξ της, ότι η ομάδα μας ε, συμφωνεί ε, στην ε, περαιτέρω βελτίωση του τελωνιακού κώδικα και πρέπει να συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας για καλύτερη συνεργασία και λειτουργία των τελωνιακών αρχών. Και επίσης θα πρέπει να ανταποκριθούμε στη βασική ανάγκη εναρμόνισης των ελέγχων που διενεργούν οι τελωνιακές αρχές οι εθνικές τελωνιακές αρχές αλλά και οι αρχές διαχείρισης των λιμένων γνωρίζουν αυτό που σημαίνει δηλαδή ότι ορισμένοι ε, μεταφορείς επιλέγουν λιμένες ε, με λιγότερους ελέγχους και αυτό βέβαια οδηγεί σε στρεβλώσεις ε, στις ροέ ε, των ε, αγαθών, ε, πράγμα το οποίο βέβαια έχει και δημοσιονομικέ επιπτώσει και δημιουργεί ένα γενικότερο αρνητικό πλαίσιο. Γι' αυτό θεωρούμε ενδιαφέρουσα την πρόταση των Πρασίνων να αξιολογηθεί ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος αυτής της στρέβλωσης αυτής, δηλαδή ανακατεύθυνση των εμπορικών ροών. Για να επιτευχθεί λοιπόν αυτόν, θεωρούμε ότι θα πρέπει να εναρμονιστούν τα πρότυπα ελέγχου των τελωνιακών αρχών και επίση θεωρούμε ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί μια κοινή αρμόδια αρχή, η οποία ακριβώ θα είναι αρμόδια για την είσοδο, ειδικότερα μέσω από το λιμένο των εμπορικών αγαθών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, και ε, για να ανταποκριθεί στι ε, υποχρεώσει τη αυτή μια υπηρεσία προτείνει η δική μου ομάδα την ε, δημιουργία νέων δικτών για την αξιολόγηση των σχετικών δράσεων. Από την άλλη πλευρά η ολοκλήρωση τη Τελωνιακή Ένωση και διασφάλιση τη ίση μεταχείριση όσων εισέρχονται στου λιτουμένου μα σημαίνει ακριβώ ότι θα πρέπει να υπάρξει εναρμόνιση των σχετικών κανόνων. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε δηλαδή ότι η εναρμόνιση των κυρώσεων παίζει σημαντικό ρόλο όπω έχει ζητηθεί και από κάποια κράτη-μέλη ό,τι αφορά την ε, στρέβλωση του εμπορίου, θεωρούμε πω η αρχική διατύπωση τη έκθεση εστιάζει ειδικότερα ε, στην καταπολέμηση των παραποιημένων ε, προϊόντων. Αλλά θεωρούμε ότι θα πρέπει να τονίσουμε και άλλα ζητήματα που είναι που σχετίζονται με το παράνομο εμπόριο και παράδειγμα όπως η τρομοκρατία, το ξέπλυμα βρωμικού χρήματος, η εμπορία αγρονιδών και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν θα κάνουμε κάποιες τροπολογίες ε, από την δική μας ε, ε, πλευρά ούτως ώστε να υπάρξει αποτελεσματικότερη καταπολέμηση των παράνομων χρηματοοικονομικών ροών και θεωρούμε πως αυτή η προσπάθεια θα πρέπει να γίνει σε δύο επίπεδα και μέσω του καλύτερου συντονισμού και της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ τελωνιακών αρχών αλλά και διαφορετικών αρμοδίων αρχών που είναι αρμόδιες για τους γενικότερους τομείς και γι' αυτό θα υποστηρίξουμε και τις τροπολογίες για καλύτερη συνεργασία μεταξύ των διάφορων συναρμόδιων υπηρεσιών της ε, Επιτροπής και αφετέρου ε, στο επίπεδο της εξωτερικής επιτυχής ενισχύοντα τη συνεργασία με τρίτες χώρε τόσο στο επίπεδο των ελληνικών αρχών όσο και σε άλλα διοικητικά επίπεδα. Θα πρέπει να συνεχίσουμε την ανάπτυξη στρατηγικών οι οποίε προωθούν την προστασία και την, ανάπτυξη των, ε, και την προστασία των ε, δικαιωμάτων πνευματική ιδιοκτησία και στις ε, τρίτε χώρε. και θεωρούμε πω θα πρέπει να δημιουργηθεί και να εδρεωθεί ένα, σταδιακά ένα σύστημα γεωγραφικών ενδύσεων των αγροτικών προϊόντων όπω έχει ήδη προταθεί από ορισμένα μέρη. Θεωρούμε λοιπόν καταληκτικά ε, από την πλευρά τη δική μα ομάδα ότι χρειάζεται όχι μόνο καλύτερο συντονισμό και συνεργασία μεταξύ των τελωνιακών αρχών και περισσότερη αναρμόνιση των σχετικών ε, κανόνων, των ελέγχων, των κυρώσεων. Αυτό θα αποτρέψει τη δημιουργία στρεβλώσεων στου λιμένε εισαγωγή στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση και θα διασφαλίσει ότι όλα τα προϊόντα που εισέρχονται στην επικράτηση τη Ευρωπαϊκή Ένωση συμμορφούνται με τα σχετικά κριτήρια και μπορείτε να είστε σίγουροι ότι θα συμμετάσχουμε μικροδομητικά στη σχετική προσπάθεια. Thank you, Chairman. Um... Ε, τους ε, Το νέο σύστημα που θέλουμε να δημιουργήσουμε σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να δημιουργήσει εμπόδια στο εμπόριο, ε, χρονικές καθυστερήσεις και ούτω καθεξής. Και αυτό μας απασχολεί όταν εξετάζουμε την σχετική έκθεση για την διευκόλυνση του εμπόριου. Ε, υπάρχουν πολύ περίπλοκοι κανόνε τελωνιακών ελέγχων και διαφορετικά συστήματα ε, κυρώσεων που εφαρμόζονται από τι διαφορετικέ αρχέ, πράγμα το οποίο ε, μπορεί να αποτελέσει μεγάλο βάρος για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και βέβαια αποτελεί και επιβάρηση ε, σε επίπεδο προϋπολογισμού. Άρα λοιπόν θεωρούμε πως θα πρέπει να εξετάσουμε τις δυνατότητες συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών και των εμπλεκόμενων φορέων τόσο ώστε να αντιμετωπίσουμε τα κοινά που υπάρχουν στο επίπεδο των τελωνιακών ελέγχων και επίσης θα πρέπει να υποστηρίξουμε τα κράτη-μέλη στο επίπεδο της εφαρμογής ε, απλουστεύσεων των ε, τελωνιακών κανόνων. Και εδώ νομίζω πως θα πρέπει να συνεργαστούμε και πιο εντατικά με τον ιδιωτικό τομέα γιατί και εκείνο ε, ε, ε, επιθυμεί να υπάρξει μια βελτίωση. Θα πρέπει δηλαδή να συνεργαστούμε με αυτού του φορεί σε ό,τι αφορά και ε, το παράνομο εμπόριο συμπεριλαμβανομένη τη εμπορία άγριων ειδών. Θα πρέπει η Επιτροπή επίσης να αξιολογήσει αξιοποιήσει πολύ ευρύτερα τον, την έννοια των εγκεκριμένων οικονομικών εφορέων και επίσης θα πρέπει αφενός να διευκολυνθεί το εμπόριο, αλλά από την άλλη πλευρά να διατηρηθούν οι πολύ αυστηροί ε, κανόνες ε, συμμόρφωσης, έτσι ώστε οι ε, οι επιχειρήσει που δραστηριοποιούνται στι τρίτε χώρε να συμμορφούνται με του σχετικού κανόνε. Δεν είμαστε πεπισμένοι ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί μια κοινή αρμόδια αρχή στο επίπεδο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίση, θεωρούμε ε, ότι θα πρέπει να επανεξετάσουμε το ζήτημα της οδηγίας για τις ακυρώσεις. Θα πρέπει δηλαδή να, υπάρχει κοινό, να υπάρχουν κοινοί ε, εδώ, ε, κοινοί κανόνες ε, για όσους για παράδειγμα παραβιάζουν τους σχετικούς κανόνες, αλλά θεωρούμε πως ήδη υπάρχουν τέτοιου είδους διατάξεις στον τελωνιακό κώδικα που προβλέπουν δηλαδή ότι σε επίπεδο κρατών μελών θα πρέπει να ληφθούν ακριβώς τέτοιου είδους αναλογικά μέτρα. Επίσης θα πρέπει να εξετάσουμε το πώς αξιοποιείται το ηλεκτρονικό εμπόριο προκειμένου να γίνει εισαγωγή παραβιάζοντας παραποιημένων αγαθών ε, στην ε, επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επίσης θα πρέπει να δούμε πώς αξιολογικούμε τους σχετικούς ε, κινδύνους, ειδικότερα στο επίπεδο δηλαδή της καταπολέμησης των παραποιημένων προϊόντων. Πάντως αυτό που πραγματικά είμαστε πεπισμένοι ότι θα πρέπει να κάνουμε είναι ότι θα πρέπει να συνεργαστούμε καλύτερα με τους συναρμόδιους φορείς, με τον ιδιωτικό τομέα και αναμένουμε και εμείς με ενδιαφέρον τις συζητήσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Για την δεν βλέπω να υπάρχει κάποιος εκπρόσωπος. Επομένως, στρέφομαι προς την ΚΟΕ. Κύριε Σόλτς, ευχαριστώ πολύ. Πολύ σύντομα, διότι η κυρία Μινόρη Σιώδης μας είναι άρρωστη και δεν μπόρεσε να έρθει σήμερα. Οπότε εγώ μίλησα απλά λίγο μαζί της τηλεφωνικά για να σας πω την ε, δική μας τάση. Συμμεριζόμαστε την ε, προσέγγιση της εισηγήτριας και την υποστηρίζουμε. συμφωνούμε ότι η συνεργασία μεταξύ των γενικών διευθύνσεων που έχουν αρμοδιότητα ε, στα τελωνικά ζητήματα και μεταξύ των τελωνικών αρχών των κρατών πρέπει να ενισχυθεί. Συμφωνούμε και εμείς ότι θα πρέπει να υπάρχει ανταλλαγή προφοριών με διαφάνεια. Τέλος, συμφωνούμε επίσης ότι θα πρέπει ε, οι τελωνικές αρχές να επικεντρώνονται και των 28 κρατών μελών να επικεντρώνονται στην συνεργασία με τις τελωνιακές αρχές των τρίτων χωρών. Και αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο αφορά μια σειρά από άλλα θέματα επίσης, ε, οριζόντια, όπως είναι η καταπολέμηση διαφθοράς, ε, η καταπολέμηση των ανισοτήτων και της κοινωνικής αδικίας ε, και θα ήθελα και αυτά τα στοιχεία να ε, ενταχθούν στην ε, έκθεση της Επιτροπής μας. Ο Πρόεδρος, εκτός μικροφώνου. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ και την εισηγήτρια. Νομίζω ότι η συνεργασία είναι πολύ επικοδομητική μαζί της. Οι τροπολογίες μας επικεντρώνονται σε τρεις προσεγγίσεις. Ζητούμε καλύτερη συνεργασία των τελωνιακών αρχών στην καταπολέμηση κατά των ε, ε, παράνομων ε, χρηματοοικονομικών ροών. Δεύτερο θέμα, το οποίο ανέφερε ήδη η συγγήτρια και το ανέφερε και ο κύριος Σούστερ, θέλουμε να ευαισθητοποιήσουμε γύρω από τα ζητήματα του περιβάλλοντος που σχετίζονται με την επιλογή από τους εισαγωγείς της ευκολότερης πύλης εισόδου. Αυτό ε, δημιουργεί περιτές ε, οδικές μεταφορές και τεράστιο όγκο ε, αερίων του θερμοκηπίου ενώ επιβαρύνει και την υποδομή μόνο και μόνο προκειμένου να αποφεύγονται συγκεκριμένοι λιμένες. Τρίτο σημείο είναι ότι πιστεύουμε ότι χρειάζεται εξαίρετη εκπαίδευση των τελωνιακών, των εργαζομένων των τελωνιακών αρχών όσον αφορά την επιμέλεια, όπως είναι για παράδειγμα η νόμιμη ξυλία ή ο σεβασμός των εργασιακών ε, ε, συνθήκων και δικαιωμάτων στον τομέα των ενδυμάτων. Συμμεριζόμαστε τις ανησυχίες της συγγήτριας και από αυτή την άποψη ε, προσβλέπουμε σε μια επικοδομητική συνεργασία μαζί της στην πορεία κατάρτισης του κειμένου. Το ΙΕΝΕΦ e λέει ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρόκειται για ένα θέμα το οποίο μας αφαιρά άμεσα, αφορά την ε, κυριαρχία των κρατών και εμείς είμαστε υπέρ μιας ένωσης συνεργασίας μεταξύ κρατών, επομένως εναρμόνιση και σε φορολογικό και σε τελωνιακό επίπεδο θεωρούμε ότι σήμερα δεν υπάρχει δυνατότητα εναρμόνισης ε, και τη σύσταση ε, κεντρικών οργανισμών. Εμείς είμαστε υπέρ του σεβασμού της αρχής της επικουρικότητας, η οποία εφαρμόζεται κατεξοχήν, διότι για μας ε, τα τελωνία εξαρτώνται απευθεία από το Υπουργείο Οικονομικών. Και διαπιστώσαμε στη Γαλλία, με όλη την κρίση που είχαμε τα δύο τελευταία χρόνια με την τρομοκρατία, ότι τα τελωνία δεν ήταν τόσο αποτελεσματικά αποτελεσματική όταν ανήκε σε άλλους οργανισμούς από ότι όταν ήταν ανεξάρτητη. Ε, θεωρούμε λοιπόν ότι σήμερα η ανάγκη είναι να υπάρχει μεγαλύτερη συνεργασία και όχι εναρμόνιση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Και τώρα να δώσουμε το λόγο στα μέλη. Υπάρχει κάποιος ο οποίος θέλει το λόγο. Παρακαλώ. Ναι. Κύριε Πρόεδρε, για να προσθέσω και κάτι στα όσα είπε ο κύριος Μπούχνερ ήδη εκ μέρου των Πρασίνων, θα ήθελα να επισημάνω και εδώ θα ήθελα να ε, ρωτήσω και την εισηγήτρια αλλά και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι τα τελωνία δεν είναι απλώς πάρα πολύ σημαντικός ε, ε κόμβος φυσικών ε, εμπορικών ροών, αλλά είναι και κόμβος ροών πληροφοριών για την αλυσίδα διανομής. Και Έχω ακούσει τον ισχυρισμό ότι στις Ηνωμένε Πολιτείε οι τελωνιακέ πληροφορίε, διατίθεται πολύ πιο εύκολα δημοσίως από ό,τι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και γιατί θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό όσον αφορά την αυξανόμενη ζήτηση και την ανάγκη να υπάρχει διαφάνεια στις αληθίδες διανομής. Ε, πιστεύω ότι θα πρέπει και εμείς να δούμε μήπως θα έπρεπε να προτρέψουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, να δει κατά πόσο θα μπορούσε να υπάρχει δημόσια πρόσβαση τελωνιακών πληροφοριών. Βεβαίως μπορεί να υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί αλλά νομίζω ότι υπάρχουν εξαιρετικά μέσα να ε, αντιμετωπίσουμε το θέμα της διαφάνειας της αληθινής διανομής, ιδίω για εισαγωγές από χώρε οι οποίες δεν ε, σέβονται βασικούς εργασιακούς ε, και περιβαλλοντικούς κανόνες και κανόνες διαχείριση. διαχείρισης. Ερώτηση λοιπόν προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μπορείτε να το λάβετε υπόψη και θεωρείτε ότι θα μπορούσε να συμπεριληφθεί σε αυτή την πρόταση. Ευχαριστώ πολύ για τις παρατηρήσεις να ρωτήσω και πάλι στους συναδέλφους αν υπάρχει κάποιος άλλος ο οποίος θέλει να κάνει κάποια παρατήρηση. Όχι, η Κομισιόν λοιπόν. Παρακαλώ. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Εκ μέρους της Κομισιόν θα ήθελα να δάξω την ευκαιρία για να ευχαριστήσω ε, την Επιτροπή σας για αυτή την πολύ σημαντική πρωτοβουλία για την αξιολόγηση των εξωτερικών παραμέτρων της επίδοσης και της λειτουργίας των τελευταίων αρχών. Εμείς εξακολουθούμε να ε, εξετάζουμε ακόμη τις τροπολογίες αλλά και τα σχόλια που ακούστηκαν σήμερα ε, και θα τοποθετηθούμε όταν υποβληθεί το σχέδιο έκθεσης, το οριστικό σχέδιο έκθεσης και προσβλέπω στην περαιτέρω συζήτηση και συνεργασία με την Επιτροπή σας ε, επί του συγκεκριμένου θέματος. Ευχαριστώ. Ωραία, λέει ο Πρόεδρος. Συνάδελφε, Χάουταλα είμαι. Είμαι η κυρία Χάουταλα, αν δεν γνωριζόμαστε. Εν πάση περιπτώσει, Νομίζω ότι η ερώτησή μου ήταν καλά διατυπωμένη και σαφής. Οπότε θα ήθελα να λάβω μία τουλάχιστον σε αδρές γραμμές απάντηση της Κομισιόν, η οποία ήταν πάρα πάρα πολύ σύντομη, γιατί νομίζω ότι αυτός είναι και ο δικός μας ρόλος, να ρωτάμε, ε, να θέτουμε ερωτήσεις στην Κομισιόν και εκείνη να μας απαντά. Πρόεδρος, δίκιο έχετε σε αυτό που λέτε. Ε, και εγώ θα ήθελα να ξαναστραφώ στην Κομισιόν ε, και να, να επιμείνω. Έχετε ενδεχομένως κάποιες ουσιώδεις πληροφορίες να υποβάλλετε σε σχέση με τα όσα ακούστηκαν από τα μέλη της Επιτροπής μας. Αν ναι, παρακαλώ μοιραστείτε τις μαζί μας. Ευχαριστώ πολύ. Εξ όσων γνωρίζω, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή πρόταση προκειμένου να σας απαντήσω. Ε, δεν έχουμε αυτή τη στιγμή τουλάχιστον σκοπό ε, να ε, αντιγράψουμε κατά κάποιο τρόπο το αμερικανικό μοντέλο. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τέτοια πρόταση. Αυτό μπορώ να σας πω αυτή τη στιγμή. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι η Κομισιόν αρνείται να εξετάσει ενδεχομένως μια τέτοια πρόταση, μια τέτοια προοπτική. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τίποτα σχετικό και γι' αυτόν τον λόγο δεν έχω και τίποτα παραπάνω να σας πω. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Και στρέφομαι ξανά στην εισηγήτριά μας για το κλείσιμο της ε, συζήτησης μας. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα είμαι πολύ σύντομη. Νομίζω ότι και από αυτά που ακούσαμε ε, διαπιστώνουμε ότι όλοι θέλουμε να, βρεθούμε, να βρούμε ένα κοινό κείμενο, επομένως δεν νομίζω ότι θα καθυστερήσουμε πολύ. Θα υπάρξει μια πρώτη συνάντηση, ελπίζω ήδη από την επόμενη εβδομάδα. Για τις πληροφορίες συμφωνώ και εγώ απολύτως ε, με τα όσα είπε η κυρία Χάουταλα. Και σίγουρα υπάρχουν κάποιες τροπολογίες που προς αυτό ε, σκοπεύουν. Ε, ελπίζω λοιπόν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να υπάρξει συγκεκριμένο αίτημα ε, και από εκεί και πέρα να αναλάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να δώσει κάποια συνέχεια. Ελπίζω ήδη από την επόμενη εβδομάδα να μπορέσουμε να συναντηθούμε. Θα φροντίσω να σας ε, προτείνω κάποια ημερομηνία το συντομότερο δυνατόν και ευχαριστώ πολύ για τη συνεισφορά σας και πάλι. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα συζήτηση για τις συμβαστικές τροπολογίες θα γίνει στη συνέχεια, διότι θα ψηφίσουμε στην επόμενη ε, συνεδρία της Επιτροπής μας και θα προσπαθήσω βεβαίως να δούμε και τι μπορούμε να κάνουμε για τους δισταγμούς που εξέφρασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σήμερα. Νομίζω ότι είναι ασυνήθιστο κάτι τέτοιο και η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίων ε, έχει μάθει να παίρνει απαντήσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ. Επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη, σημείο υπαριθμών 7. Θέσπιση κανόνων για τη διάθεση λιπασμάτων με σήμανση CE στην αγορά. Πρόκειται για γνωμοδότηση. Και εδώ και σε αρκετές επιτροπές έχουν γίνει αρκετές συζητήσεις για τον κανονισμό για τα φυτοφάρμακα και τα λοιπάσματα. Θα ήθελα να υπενθυμίσω στα μέλη ότι και στο θέμα αυτό, όπως και στο προηγούμενο θέμα, θα πρέπει να προσέξουμε και το ε, ε, πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου. Να δώσουμε το λόγο στο συντάκτη της γνωμοδότησης, ο κύριος Μπαλές από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρόκειται για ένα πολύ περίπλοκο ζήτημα, οπότε εκ των προτέρων σας ζητώ συγγνώμη και σας προειδοποιώ ότι θα επεκταθώ λίγο σε με αυτό το ζήτημα. Είναι τρίτη φορά που συζητάμε αυτό το ζήτημα ε, και έχω αναφέρει και τις ανησυχίες εμπορικού χαρακτήρα. Ε, υπάρχουν ε, κάποια ερωτήματα που έχουν τεθεί καταρχήν σε ό,τι αφορά το ζήτημα αρμοδιότητας της δικής μας Επιτροπής της αλλά δεν μπορώ να φανταστώ ότι σε σχέση με ένα τόσο σημαντικό για εμπορικά ζητήματα φάκελο ε, να εξαιρεθεί η Επιτροπή μας. Ε, και για να σας το πω πολύ απλά, συζητούμε όρια σε ό,τι αφορά εισαγωγές εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όρια τα οποία ουσιαστικά ε, καταστρέψουν ουσιαστικά τις εξαγωγικές αγορές των βορειοαφρικανικών χωρών και αλλαγές οι οποίες θα δημιουργήσουν και διαφορές σε επίπεδο δηλαδή Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίων και για αλλαγέ οι οποίε θα καταστήσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση εξαρτημένη από τι αγωγέ. Οπότε δεν έχουμε λόγο σύντα, δεν νομίζω ότι δεν έχουμε λόγο. Οπότε ε, νομίζω πω και οι περισσότεροι από εσά θα συμφωνήσετε μαζί μου, ακόμα και αν δεν συμφωνείτε μαζί μου ε, επί του ότι δηλαδή ε, θα πρέπει να συμμετάσχουμε ενεργά στη διαμόρφωση των γενικότερων παραμέτρων αυτού του κανονισμού γιατί αυτό είναι και ο ρόλος μας εδώ εντός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτό καλούμαστε να κάνουμε και εγώ σε καμία περίπτωση δεν θα παραμείνω σε βουλός. Ελπίζω και εσείς ε, να με βοηθήσετε και να με υποστηρίξετε σε αυτή την προσπάθεια. Τώρα, να περάσω στην ουσία αυτού του φακέλου. Κατά την τελευταία μα συνεδρίαση είχα αναφερθεί σε μια σειρά από ζητήματα τα οποία πηγάζουν από το ίδιο βασικό ε, ζήτημα. Δηλαδή, η Επιτροπή προτείνει συγκεκριμένα επίπεδα καδμίου σε λοιπάσματα, ε, τα οποία όμω είναι ουσιαστικά μη ρεαλιστικά, δεν μπορούν να επιτευχθούν από, την, από τον κλάδο και γι' αυτό το λόγο αναφέρθηκαν τέσσερα ζητήματα. Η, καταρχήν η εξάρτηση από τι εισαγωγέ. Δηλαδή, η Ευρωπαϊκή Ένωση εξαρτάται έως και κατά 90% από τις αγωγές φωσφορίτη. Παρότι δηλαδή ο φωσφορίτης ε, θεωρείται ως κρίσιμη πρώτη, critical raw material, η Επιτροπή δεν έχει κάνει πολλά ε, προκειμένου να ανοίξουν περισσότερες ε, προμήθειες από την αλλοδαπή. Έτσι ε, οι περιορισμένες ε, προμήθειες ε, που υπάρχουν θα γίνουν τώρα διαθέσιμες για όλου και αυτό θα δημιουργήσει ακόμα μεγαλύτερες δυσκολίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση να λαμβάνει καθαρό φωσφορίτη και θα είναι υποχρεωμένη να προμηθεύεται αυτό το φωσφορίτη από συγκεκριμένες επιχειρήσεις. Μετά, δεύτερο ζήτημα, η μόνη επιστημονική μελέτη η οποία υποστηρίζει τα όρια που προτείνει η Επιτροπή αναφέρεται σε 80 80 ε, μιλιγκράμμ, το οποίο βέβαια ε, υποτίθεται πως αποκρίνεται στη συσσόρευση καθμίου στο έδαφος. Εάν λοιπόν σε αυτό το όριο των 80 μιλιγκράμμ δεν δημιουργήσει συσσόρευση του καρμίου στο επέδαφο, τότε γιατί η Επιτροπή έχει χρησιμοποιήσει τα όρια των 60, 40, 20 μιλιγκράν. Δεν έχω βρει δηλαδή κάπου αλλού κάποια θεμελίωση αυτή τη άποψη και έχω θέσει αυτό το ερώτημα στην Επιτροπή εδώ και ένα χρόνο. Ε, πέραν αυτού, ε, εδώ ε, τα όρια που προτείνει η Επιτροπή δεν είναι μέσο όρο περιεκτικότητα. Αναφέρεται σε ανώτατα όρια η πρόταση τη Επιτροπή σε καδμίου στα λοιπάσματα. Από εκεί και μετά, ε, διαφορέ οι οποίε θα πρέπει να θα τεθούν σε επίπεδο. Ε, ΠΟΕ. Είναι πιθανό οι ε, εν λόγω προτάσει να μην συμμορφώνεται με τους κανόνες του ΠΟΕ, οπότε αυτό μπορεί να ε, δημιουργήσει ακριβώς ένα, να ξεκινήσει μια διαφορά την οποία τελικά θα χάσει η Ευρωπαϊκή Ένωση ακριβώς επειδή δεν υπάρχει κατάλληλη επιστημονική βάση που να θεμελιώνει αυτή την, ε, αυτά τα προτινόμενα όρια καρμίου. Από εκεί και μετά ε, υπάρχει το σύστημα του εκβιασμού από, από συγκεκριμένες ε, χώρες, δηλαδή καθώς υπάρχουν χώρε οι οποίε εξάγουν το κάδμιο προ την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά είναι ανταγωνιστέ τη σε ό,τι αφορά τα έτοιμα λιπάσματα, τα έτοιμα προϊόντα λοιπόν, τα τελικά προϊόντα λίπανση, είναι πιθανό οι σχετικοί εξαγωγείς να αξιοποιήσουν και να καταχραστούν τη θέση τους. Και αυτό συνέβη πριν από κάποια χρόνια όταν μια επιχείρηση χρειάστηκε να ουσιαστικά δωροδοκίσει δύο ε, παραγωγούς της Ρωσίας ώστε να μπορέσει να έχει πρόσβαση ακριβώς στις ε, προμήθειες ε, καθαρού φωσφορίτη. Αυτό λοιπόν αποτελεί μια πραγματικότητα. Θέλουμε πραγματικά, ρωτάω, να εξαρτώμαστε από εισαγωγέ από ξένε χώρε φωσφορίτη. Ε, ε, και εδώ αναφερόμαστε βέβαια για την ασφάλεια των τροφίμων. Ε, οπότε, ναι, είμαι και εγώ υπέρ του να κινηθούμε προς χαμηλότερες περιεκτικότητες πηγές καδμίου, να βρούμε σε διαδικασίες αποκαδμίωση αλλά και θα πρέπει και να προωθήσουμε και την κυκλική οικονομία σε αυτή τη βιομηχανία, έτσι ώστε να μειώσουμε την εξάρτησή μα από τι ε, εισαγωγέ από ξένε χώρε. Αλλά όλα αυτά θα πρέπει να γίνουν με τρόπο ο οποίο θα διασφαλίσει την ανάπτυξη και την επιβίωση του κλάδου των ε, λιβασμάτων. Δεν θα πρέπει δηλαδή στο πλαίσιο αυτή τη διαδικασία να καταδικάσουμε σε θάνατο τον ελόγο κλάδο. Οπότε ε, Ε, παρότι δεν μπορώ να αναφερθώ στα συγκεκριμένα όρια τα οποία δόθηκα μόνο στην ένδυση ό,τι αφορά το παράτημα της πρότασης, αλλά ε, υπάρχουν ε, ε δύο συγκεκριμένε προτάσεις που γίνονται για να ε, διορθώσουμε αυτή την κατάσταση. Παρότι λοιπόν το πρώτο παράτημα του κανονισμού προτείνει ανώτατα όρια, εγώ προτείνω από τη δική μου πλευρά με βάση και μια πρόσφατη επιστημονική μελέτη για τη συσσόρευση κατμίου, να ισχύει το όριο των 80 μιλιγκράν κατά μέσο ώρα από την πλευρά των ε, προμηθευτών όπως προτείνεται από τον ε, ε, καθηγητή Σμόλτερς. Δεύτερο, με βάση ακριβώς τις, την εξάρτηση από τις εγωγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης προτείνω ένα μηχανισμό λήψης ή μάλλον χορήγησης μιας προσωρινής απόκλησης για παραγωγούς οι οποίοι δυσκολεύονται ακριβώς να βρουν πηγές ε, προμήθειας ε, καδμίου και αυτό το σύστημα θα ε, βασίζεται σε εκθέσεις σε προϊόντα οι οποίες θα υποβάλλονται και στην Επιτροπή και στο Κοινοβούλιο και από εκθέσεις σε ό,τι αφορά τις προσπάθειες που γίνονται ακριβώς για την λήψη από πηγές χαμηλής περιεκτικότητας καδμίου από, μέσω της αποκαδμίωσης επίσης και μέσω της κυκλικής οικονομίας τέλος ε, προτείνω ε, ακριβώς για να αποφύγουμε τη δημιουργία διαφορών σε επίπεδο ε, ΠΟΕ ένα δικό μας ε, μηχανισμό ο οποίος θα μας επιτρέψει να αποφύγουμε μια τέτοια ε, κατάσταση. Τέλος, επειδή υπάρχει ο κίνδυνος ακριβώς να καταχραστούν αυτά τα νέα όρια οι εξαγωγής των τρίτων χωρών έτσι ώστε δηλαδή να αξιοποιήσουν καλύτερα την αποκλειστική πρόσβαση που θα έχουν σε καθαρό φωσφορίτη και κατά συνέπεια ε, το μονοπόλιο τρόπο που θα έχουν σε ό,τι αφορά τα τελικά προϊόντα λίπανσης, ε, προτείνουμε ε, στην Επιτροπή να παρέμβει και να αποθαρρύνει τις τρίτες χώρες έτσι ώστε να μην καταχαστούμε αυτόν τον τρόπο την προνομιακή τους θέση τέλος λαμβάνοντας υπόψη τα πεπερασμένα από θέματα που υπάρχουν στην παγκόσμια αγορά του καθαρού φωσφορίτη, ζήτησα από την Επιτροπή να προετοιμάσει μια σχετική έκθεση και να αναφέρει ε, ε, τι περιπτώσει χωρών οι οποίε συσσωρεύουν ουσιαστικά αυτή την πολύ κρίσιμη πρώτη ύλη για τον εαυτό του, έτσι ώστε να αναλάβει στη συνέχεια η Επιτροπή δράση εναντίον αυτών των χωρών. Αυτά λοιπόν είναι τα βασικά στοιχεία τη δική μου ε, πρόταση και αναμένω τώρα με ενδιαφέρον τα σχόλιά σα. Ευχαριστώ για όλα αυτά και περνάμε στους σκιώδεις. Εκ μέρους των σοσιαλιστών, ο κύριος Αντριώ. Ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, αγαπητοί συνάδελφοι και κύριε Βαλέσα, καταρχάς ε, θα ήθελα να υπενθυμίσω τη στήριξή μας ε, από πλευράς της ομάδος ε, στον κανονισμό αυτό, πολύ αναμενόμενος από το τομέα της γεωργίας και τους χρήστες φυτοφαρμάκων, και ο οποίο θα επιτρέψει να μειώσουμε την εξάρτησή μας μέσω της κυκλικής οικονομίας όπως ακούστηκε και να βελτιώσουμε και τη διάθεση οργανικών ε, προϊόντων τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά όπως όλοι γνωρίζουμε για να υπάρχει βιώσιμη γεωργία όπως ε, επιθυμούμε όλοι. Διότι η υγεία και ε, το περιβάλλον είναι σημαντικές ανησυχίες και να το, περιορίσουμε, το να περιορίσουμε συγγνώμη, ρηπογόνες ουσίες ε, στα φυτοφάρμακα είναι ο βασικός στόχος του κανονισμού αυτού. Όσον αφορά το σχέδιο γνωμοδότησης, θεωρώ ότι η ιδέα της παρακολούθησης και της υποβολής εκθέσεων είναι πάρα πολύ σημαντική, κυρίως για να δούμε τη διαθεσιμότητα σε φωσφορίτη, για να μπορούμε να δούμε αν μπορούμε να τον προμηθευτούμε. η απλούστευση για την πρακτική εφαρμογή και όταν τελειώσει και η μελέτη αντικτύπου για τις αναπτυσσόμενες χώρες ε, και περιμένουμε και την πρώτη υποβολή εκθέσεων, μπορεί να έχουμε κάποια σημαντικά στοιχεία εδώ στην Επιτροπή μας, ε, ε, τα οποία θα μπορούσαμε να υποβάλει σε άλλες αρμόδιες επιτροπές. Έχω όμως κάποια ερωτηματικά κατά πόσον είναι εφικτό ή αρμόζει σε αυτόν τον κανονισμό να αναφέρουμε κάποια πράγματα, όπως για παράδειγμα τις κυρώσεις που έχουμε στην τροπολογία 8 και 9. Επίσης, θα θέλαμε να ακούσουμε και την άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επ' αυτού. Ε, έχω και κάποιες επιφυλάξεις για κάποιες άλλες προτάσεις, όπως για παράδειγμα αυτή που αναφέρεται στην τροπολογία παριθμών 7 για την αυτόματη αναστολή ενός ε, τμήματος, ενός ευρωπαϊκού ε, κανονισμού όταν ένα κράτος υποβάλλει ένσταση στον ΠΟΕ. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει de facto εξουσία σε τρίτες χώρες, αν κατάλαβα καλά, να ε, ζητούν αναστολή εσωτερικού κανονισμού και αυτό αποτελεί ουσιαστικά και πρόσκληση για να το υλοποιήσουν. Ε, οποιοδήποτε και αν είναι το θέμα, εγώ δεν μπορώ να προσυπογράψω τέτοια κίνηση. Το δημιουργήσουμε εμείς μόνοι μα υποψίες στο δίκαιό μας, ε, νομίζω ότι δεν συνάδει με το ρόλο του νομοθέτη. Τουλάχιστον έτσι αντιλαμβάνομαι εγώ τις προτάσεις αυτές. Όσον αφορά το θέμα του, των κατοφλίων, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για την γνωμοδότησή μας. Αυτή τη στιγμή που συζητάμε δεν ξέρουμε ακριβώ ποια θα είναι τα όρια, διότι οι συνάδελφοι της Επιτροπής Περιβάλλοντος και των ε, Εθνικών ε, Κοινοβουλίων που θα καθορίσουν τα τελικά μέτρα. Και αυτό φυσικά δημιουργεί και πάλι ερωτηματικά για το τι αρμοδιότητα έχουμε εμείς εδώ ως Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Για να ολοκληρώσω, νομίζω ότι θα πρέπει να βρούμε ένα κατάλληλο τρόπο να ε, θέσουμε τις ανησυχίε μας στις αρμόδιες επιτροπές του Κοινοβουλίου και νομίζω ότι η Γραμματεία θα πρέπει να μας δώσει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο επί το οποίο θα πρέπει να εργαστούμε συλλογικά. Σας ευχαριστώ πολύ. Uh, Ευχαριστώ πολύ. Από τους συντηρητικούς, η κυρία Μακλάρν. Ναι. Εκπροσωπώ τον κύριο Πιέκα. Το ECR υποστηρίζει πλήρως τις θέσεις του εισηγητή για τον νέο κανονισμό. Δεν έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση φωσφορίτη, επομένως πρέπει να τον εισάγουμε, γι' αυτό και εξαρτόμαστε από τις ε, τρίτες χώρες. Από αυτήν την, ε, σε, αυτήν, σε αυτόν τον τομέα αυτού του πολύ της, αυτής της πολύ κρίσιμης ε, πρώτης ύλης. Τα όρια ε, καταλήπων και ρηπογόνων ουσιών ε, υπερβαίνουν τις ε, ικανότητες που μπορούν να και θεσπίζουν κανόνες που δεν μπορούν να τηρήσουν οι περισσότεροι παραγωγοί. Το μεγαλύτερο μέρος του φωσφορίτη προέρχεται από χώρες όπως η Ρωσία, η Συρία και το Μαρόκο. Αυτό σημαίνει ότι ε, η Ευρώπη θα καταστεί εξαρτημένη. Ε, θα ε, χαθούν δε μέσω του κανονισμού αυτού και τα ωφέλη του, της εναρμόνισης ενώ θα χαθούν και οφέλη ε, όπως για παράδειγμα η πρόσβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αποθέματα της Νορβηγίας και έτσι θα ενισχυθεί η θέση της Ρωσίας. Ευχαριστώ. Άλντε δεν υπάρχει εκπρόσωπος, οπότε στρέφομαι στον κύριο Σόλτ από την ΚΟΥΕ. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ε, και σε αυτό το θέμα η ισχυρότητα μας λείπει. Θέλω να τονίσω ωστόσο ότι έχουμε ε, λάβει υπόψη μας την πρόταση της Κομισιόν και γνωρίζουμε όλοι ότι μιλούμε για ένα πάρα πολύ ευαίσθητο θέμα. Μιλούμε για τη δημόσια υγεία, υγεία για την ιατρική περίθαλψη, ε, είναι ένα θέμα που αφορά τη γεωργία, το περιβάλλον. Πρόκειται λοιπόν για ένα ε, ζήτημα ε, που άπτεται και της επίτευξης των στόχων για τη βιώσιμη ανάπτυξη ε, τόσο από πλευρά Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και στο πλαίσιο του ΟΗΕ στο χρονοδιάγραμμα που έχει συμφωνηθεί. Γι' αυτό και χαιρετίζουμε την ε, προσέγγιση που έχει υιοθετηθεί σε σχέση με, με, τους, ε, με τα λοιπάσματα και την κατάταξή τους βάση κινδύνου. Έχω και μια ερώτηση προς τον συζητητή, γιατί εξήγησε επιμακρών τη δική του θέση, αλλά και προς την Κομισιόν είστε έτοιμοι να αποδεχθείτε περαιτέρω μείωση των ορίων καδμίου στα λοιπάσματα για λόγους κινδύνου ε, για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον. Εμείς επίσης προτείνουμε ότι θα, να, ε, τη θέσπιση μάλλον δεσμευτικών μέσων και εργαλείων για να παρακολουθείτε η εφαρμογή και η τήρηση των ορίων αυτών σε όλη την κλίμακα του συστήματος. Κύριε Βαλέσα, κατάλαβα ότι έχετε συγκεκριμένα ε, ερωτήματα. Ε, θα ήσασταν έτοιμος να εξετάσετε ή ε, ενδεχομένως να συμπεριλάβετε μια τέτοια σκέψη στη δική σας έκθεση. Κυρία Χάιντι Χάουταλα από τους Πράσινους. Ευχαριστώ. Έχω ένα σχετικό ντεζαβού. Γιατί πριν από 21 χρόνια αυτό το ε, ερώτημα τα όρια ε, του καδμίου στα φωσφορικά λιπάσματα ήταν ένα από τα ζητήματα που απασχόλησαν την διαπραγμάτευση της Σουηδίας ως προς την προσχώρηση της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί όπως αναφέρθηκε υπάρχουν χώρες ε, στη Σκανδιναβία με ε, φωσφορίτη με πολύ χαμηλή περιεκτικότητα σε κάδμιο. Γι' αυτό και προτιμώ τα φιλανδικά μακαρόνια πρέπει να σας πω, παρότι τα ιταλικά είναι εξαίρετα. Τα φιλανδικά λοιπόν είναι πολύ πιο καθαρά ε, και δεν περιέχουν κάδμιο, αυτή την τοξική ουσία. Και νομίζω ότι 20 χρόνια είναι αρκετά για να είχε διευθετηθεί αυτό το θέμα. Διότι έχουν περάσει 20 χρόνια από την προσχώρηση τη ε, χώρα μου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ακόμα δεν έχει λυθεί. Θα ήθελα να μάθω και ορισμένα περισσότερα στοιχεία σχετικά με αυτή τη μελέτη που ανέφερε ο εισηγητή. Όπου, αν κατάλαβα καλά, τα 80 μιλιγκράμμ ανά κιλό λιπάσματος δεν συσσωρεύονται στα ε, ζώντα όντα όπως οι άνθρωποι. Ε, αμφιβάλλω γι' αυτό ή εν πάση περιπτώσει είμαι αρκετά σκεπτική ως προς αυτό γιατί έχω ακούσει και αντίθετα πορίσματα άλλων ερευνών. Ε, ε, υπάρχουν βεβαίως ορισμένες εξαιρέσεις και αποκλήσεις και αυτό θα μπορούσε να ήταν μια καλή ιδέα για να λυθεί το θέμα από εδώ και πέρα. Ωστόσο πρέπει να σημειώσω ότι πρόκειται για ένα σημαντικότατο ε, ζήτημα δημόσιας ασφάλειας και δεν θα πρέπει να το εξετάζουμε μόνο από τη σκοπιά του ανταγωνισμού. Και να σας πω γιατί πιστεύω ότι η πρόταση Κομισιόν είναι καλή. Διότι Υπάρχει από την άλλη πλευρά και η πρόταση για την κυκλική οικονομία των φωσφορικών λιπασμάτων. Στη χώρα μου πριν από κάποια χρόνια διαπιστώθηκε ότι υπήρξε μια τεράστια αποθήκη, ε, αποθήκευση, συσσόρευση φωσφόρου στο υπέδαφος λόγω της χρήσης λιπασμάτων. Και αυτό βεβαίως ρηπαίνει, μολύνει και τον υδροφόρο ορίζοντα. Διαπιστώσαμε λοιπόν ότι υπάρχουν τρόποι ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης τέτοιων περιορισμένης διάθεσης πρώτων υλών, ε, ε, κάτι που ε, υλών που ενδεχομένως να μπαίνουν και στην τροφική μας αλυσίδα. Ε, πρέπει λοιπόν ε, να συγχαρώ την Κομισιόν για το γεγονός ότι έχει επιδείξει μεγάλη ευαισθησία ως προς αυτό το θέμα της κυκλικής οικονομίας. Γι' αυτό και θέλω να υποστηρίξω ε, κατά βάση την πρόταση που έχει υποβάλει η Κομισιόν. Εντάξει, ευχαριστώ. Και... Ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση αυτή. Είναι σαφές ότι η παρουσία ε, ορυκτού φωσφόρου έχει μειωθεί πάρα πολύ, κυρίως στη Γαλλία, λόγω των τιμών που εκτοξεύθηκαν και επίσης και λόγω μιας μεγαλύτερης διαφοροποίησης και πιο φυσικές πηγές. Ε, τα βιολογικά λοιπάσματα αναπτύχθηκαν στη συνέχεια και εμείς είμαστε υπέρ ενός στόχου εθνικής αυτονομίας στο θέμα αυτό. Δηλαδή να αφήσουμε σε κάθε χώρα την επιλογή να ρυθμίζει τα φυτοφάρμακά της. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ και τώρα να δώσουμε το λόγο στα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής. Η Μαρία Ρενά έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εγώ έχω δύο ε, μικρές ερωτήσεις. Ε, συμφωνώ με αυτό που είπε ο Ερίκ Αντριέ όσον αφορά την ε, ε, βοήθεια προς τις χώρες που εξάγουν ε, φωσφορούχα με μεγάλη περιεκτικότητα καθμίου ε, πώς ε, σκοπεύει να ε, δώσει και συνοδευτικά μέτρα για τις χώρες αυτές, διότι αν δεν θέλουμε να βρεθούμε ενώπιον μονοπωλίων, θα πρέπει να βοηθήσουμε αυτές τις χώρες να καθαρίζουν το φωσφορό τους, ώστε να μπορούν, τα φωσφορούχα τους, συγγνώμη, ώστε να μπορούν να συνεχίσουν τις εξαγωγές τους και να έχουμε πρόσβαση στους πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πώς σκοπεύει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να απαντήσει σε αυτό το ερώτημα. Και το Δεύτερο ερώτημα είναι δεδομένο ότι υπάρχουν συμφωνίες για εξαγωγή προϊόντων και κυρίως προϊόντων που προέρχονται από την Αφρική, γεωργικών προϊόντων για παράδειγμα, και εκεί χρησιμοποιούνται φωσφορούχα με υψηλή περιεκτικότητα καθμίου. Πώς μπορούμε να κάνουμε λοιπόν ε, αποτελεσματικούς ελέγχους και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να το συζητήσουμε συμφωνία σε ελεύθερο εμπορίου με την Αφρική εδώ στην Επιτροπή μας για να μπορέσουμε να ελέγχουμε και την ε, περιεκτικότητα καδμίου στη Γεωργία. Ευχαριστώ. Υπάρχει κάποιος άλλος ο οποίος θα ήθελε το λόγο, θέλει να σχολιάσει. Αν όχι, να δώσουμε το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε το λόγο και να ευχαριστήσω και για αυτό το σχέδιο γνωμοδότησης. Ζητώ συγγνώμη, δεν ακούσαμε όλη τη συζήτηση, γιατί ήμασταν στην Επιτροπή Περιβάλλοντος που συζητούσε ακριβώς το ίδιο θέμα. Αλλά θα σχολιάσουμε ε, λίγο τη γνωμοδότηση. Ε, να σας πω μόνο ότι κάναμε μια πολύ σύντομη προπαταρκτική ανάλυση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα ολοκληρώσουμε την ανάλυση μας ε, μόλις επισυποποιηθεί η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου βεβαίως. Ως προς την έκθεση αυτή, φαίνεται να μας λέτε ότι τα 80 μιλιγκράμμα ανά κιλό είναι ασφαλές όριο. Δεν υπάρχουν τέτοιες ενδείξεις. Το έχουμε επαναλάβει αυτό αρκετές φορές. Η παρούσα έκθεση σε κάθμιο, μέσω της διατροφής, κυρίως από τη γεωργική παραγωγή, είναι ούτως ή άλλως πάρα πολύ υψηλή και επομένως ε, ε, το γεγονός ότι δεν υπάρχει συσσόρευση δεν αποτελεί ασφαλές όριο, δεν υπάρχει αξιολόγηση αντικτύπου ε, που να υποστηρίζει μια τέτοια πρόταση και η εσωτερική μας ανάλυση αποδεικνύει ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι συμβατή με τους κανόνες του ΠΟΕ. Τώρα, όσον αφορά τις συγκεκριμένες προτάσεις της έκθεσης, φαίνεται να υπάρχει μια πρόταση να επιτρέπεται στα κράτη-μέλη να δίνονται παρεκκλήσεις από τις οριακές τιμές ε, μονομερούς, και ε, εκ μέρου όλων των υπολείπων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για μας είναι πάρα πολύ ε, περίεργη διατύπωση αυτή σε κανονισμό εναρμόνισης και όλα. Να ζητάμε να δίνονται παρεκκλήσει εξ ονόματο όλων των υπόλοιπων κρατών μελών και χωρίς τη συμμετοχή Ευρωπαϊκού Θεσμικού Οργάνου. Ε, η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ούτω ή άλλως επιτρέπει στα κράτη-μέλη να έχουν παρεκκλήσεις για να επιτρέπουν ε, μεγαλύτερη περιεκτικότητα στα φωσφορούχα, αλλά ε, χωρίς σήμανση ΣΕ. Δεν υπάρχει λοιπόν άδεια για ελεύθερη κυκλοφορία σε όλη την εσωτερική αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για μας αυτή είναι η σωστή άγουσα. Ε, θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχει ένα υψηλό ε, ποσοστό προστασία για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, για όλε δηλαδή χώρε χώρες Ευρωπαϊκή Ένωση ή τουλάχιστον τι περισσότερε και τα κράτη-μέλη που ανησυχούν για το κατά πόσον θα υπάρχουν φωσφορούχα προϊόντα για του αγρότε, μπορούν να επιτρέψουν υψηλότερα όρια, αλλά αυτά τα ε, λοιπάσματα δεν μπορούν να φέρουν σήμανση ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένω, η πρώτη μα αντίδραση είναι ότι αυτή η πρόταση μα βρίσκει ιδιαίτερα προβληματισμένους. Τώρα, το να υποχρεωθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει μέτρα για την καταπολέμηση των εμπορικών πρακτικών. Δεν θεωρούμε ότι οι κανόνες αυτοί ε, ανήκουν σε νομοθεσία εναρμόνισης. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι πρόκειται για νομοθεσία η οποία βασίζεται στο άρθρο 114 της συνθήκης, επομένως ε, εναρμόνιση των ε, ιδιωτήτων προϊόντων τα οποία μπορούν να περιέχονται, να κυκλοφορούν ελεύθερα στην ενιαία αγορά και επομένω ε, η καταπολέμηση των των εμπορικών πρακτικών και η σχετική εντολή και υποχρέωση για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θεωρούμε ότι ανήκουν σε ένα τέτοιο ε, νομοθέτημα. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ για αυτά τα σχόλια και δίνω τώρα και πάλι το λόγο στον εισηγητή μα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ποια είναι η βάση για τη συζήτηση που κάνουμε. Η μελέτη του καθηγητή Ερικ ε, του 2013. Αυτή δηλαδή χρησιμοποιήθηκε στην αξιολόγηση αντικτύπου την οποία ε, προετοίμασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αλλά αυτή η αξιολόγηση αντικτύπου ήταν αρκετά περιορισμένη, αν θέλετε, προ το εύρο ε, Δηλαδή, ουσιαστικά πολύ επιλεκτική ήταν η Επιτροπή στα όσα συμπεριέλαβε στην λόγω αξιολόγηση. Εγώ ήρθα σε επαφή με τον ε, καθηγητή Σμούλτερς ε, και εκείνος μου είπε ότι χρησιμοποιεί ε, ε τη μέση περιεκτικότητα καθμίου στο έδαφος, αλλά εδώ, στη συγκεκριμένη περίπτωση, μου είπε ξεκάθαρα ότι ανάλυσε μόνο την συγκέντρωση καδμίου στο έδαφος, δηλαδή δεν είχε αναλύσει την μεταβίβαση αυτού του καδμίου που βρίσκεται στο έδαφος στα τρόφιμα. Πάντως σας ευχαριστώ όλους για τα σχόλια που κάνατε. Θα κάνω ό,τι μπορώ προκειμένου να φτάσουμε σε μια λύση η οποία θα είναι κοινά αποδεκτή από όλους. Σε ό,τι αφορά τώρα την επιστημονική θεμελίωση της άποψής μου, εγώ έχω ζητήσει επανειλημμένα από την Επιτροπή να μου πει ποια είναι τα επίπεδα παραγωγής που αναμένουμε με αυτά τα όρια. 30 20-60% και η Επιτροπή πάντα μου λέει δεν το γνωρίζουμε ακόμα, πρέπει να το ελέγξουμε. Από εκεί και μετά η Επιτροπή επιχειρηματολογεί ότι αυτό το 20% ε, που προτείνει εκείνη στην πρότασή της αντιστοιχεί σε μια μείωση τη κέντρωση κατμιου στο εδαφος κατά 20% σε 100 χρόνια. Αλλά αν ρίξουμε μια ματιά στη μελέτη του κυρίου Σμόλτες, ε, η οποία δημοσιεύτηκε το 2013 αλλά και σε μια άλλη του, κυρίου, ε, του καθηγητή ΣΕΡ του 2015. Εκεί λοιπόν αναφέρεται ότι ήδη ε, ε, ε, αυτή τη στιγμή μειώνεται η συγκέντρωση κατά 18% στα 100 χρόνια. Και αυτό χωρίς να κάνουμε τίποτα. Δηλαδή αν θέσουμε αυτά τα όρια, τι επιτυγχάνουμε, απλά να καταστρέψουμε τον κλάδο. Τι πάμε να κάνουμε λοιπόν, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας δηλαδή, τον κλάδο. Και το τονίζω αυτό εδώ. Εγώ δεν θέλω να αποδυναμώσω τη σχετική νομοθεσία, ούτε να υπονομεύσω τα όρια που θέλουμε να θέσουμε, αλλά θέλω η λύση που θα βρούμε τελικά να λειτουργήσει στην πράξη. Δεν θέλω δηλαδή να αποφασίσουμε ότι θα έχουμε κάποια όρια ιδιαίτερα χαμηλά, γιατί πάντοτε ακούγονται καλά τα χαμηλά όρια για βαρέα μέταλλα, αλλά τελικά να οδηγηθούμε σε μια κατάσταση όπου δεν θα είναι ρεαλιστικό να εφαρμοστούν αυτά τα όρια στην πράξη. Και είναι δύσκολο να φτάσουμε εδώ σε ένα κοινό παρονομαστή, γιατί η επικοινωνία ε, που έχω αυτό τον τελευταίο χρόνο με την Επιτροπή είναι πολύ δύσκολη. Δηλαδή, όταν προβήκαμε σε ανταλλαγή απόψεων, εδώ στη δική μας Επιτροπή με την Επιτροπή, ακούσαμε κάποιες δηλώσεις από την πλευρά της, οι οποίες ουσιαστικά είναι ασφαλμένες, ε, σε κάθε περίπτωση αναλυθείς. Ε, εκείνο που εγώ θέλω να διασφαλίσω σε τελική ανάλυση είναι ότι η πρόταση που θα κάνουμε θα τα αποκρίνεται στις ελπίδες και στις προσδοκίες ε, όλων μας. Αλλά εκείνο που εγώ καλούμε να κάνω, κατά κύριο λόγο, είναι να θίξω τις, ε, τα προβλήματα που περιλαμβάνει αυτή η πρόταση κανονισμού της Επιτροπής. Οπότε ε, θα φροντίσω να λάβω επόψη μου τα σχόλια που κάνατε στις περαιτέρω τροποποίησεις αυτού του εγγράφου, αλλά πρέπει να βρούμε μία έξυπνη λύση. Πρέπει αυτή δηλαδή η λύση όταν θα οριστικοποιηθεί πραγματικά να έχει νόημα και να ε, μην υπομονεύσει το δικό μας έκλαδο. Και αύριο, κατά τη μέρια του, του μεσημεριανού γεμάτος, ε, θα γίνει μια σχετική συζήτηση, οπότε όποιος από τους συναδέλφους ενδιαφέρεται να ακούσει περισσότερα για αυτό το ε, θέμα, είναι θερμά προσκεκλημένος. Αύριο λοιπόν. Ε, το γεύμα αυτό. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ για αυτή τη συζήτηση. Ευχαριστώ και για την πρόσκληση που μας απίφθηνες για αύριο το μεσημέρι. Και με αυτό ολοκληρώνουμε την ε, σημερινή μας συζήτηση. Η προθεσμία υποβολής τροπολογιών είναι η 6η Μαρτίου στις 12 το μεσημέρι. Euh, η κυρία Ρενά, θα ήθελα να πω κάτι αντίστοιχο με αυτό που είπε η κυρία Χάουτελα προηγουμένω. Θέσαμε συγκεκριμένε ερωτήσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δεν λάβαμε απαντήσει. Μήπω θα μπορούσαν να μα απαντήσουν γραπτώ στι συγκεκριμένε ερωτήσει που θέσαμε. Ε, αντιλαμβάνομαι ότι η Επιτροπή ε, δεν έχει πάντα δυνατότητα να μας απαντά άμεσα, αλλά ε, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον αυτό το οποίο σας έθετε. Θα θέλαμε λοιπόν τουλάχιστον γραπτές απαντήσεις. Ευχαριστώ. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Ε, η Κομισιόν θέλει να απαντήσει σε αυτό το αίτημα. Ναι, φυσικά, εμείς πάντοτε υποδεχόμαστε ε, με χαρά την, ε, τις ερωτήσεις που απευθύνουν σε εμάς τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ξαναζητώ συγγνώμη που δεν μπορέσαμε να παρακολουθήσουμε τη συζήτηση από την αρχή της. Ωραία, λέει ο Πρόεδρος, και έτσι λοιπόν ολοκληρώνουμε τη συζήτηση επί του θέματος αυτού για τα λοιπάσματα. Και Πάμε στο σημείο υπαριθμών 8 της ε, σημερινής μας ε, ημερήσιας διάταξης προς ένα νέο εμπορικό πλαίσιο μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας και τον εξυγχρονισμό της Τελωνιακής Ένωσης. Έκθεση πρωτοβουλίας. Κύριος κ. Ντέβιτ Μπορέλη είναι ο εισηγητής μας. Και θα θυμάστε συνάδελφοι ότι στις 21 Δεκεμβρίου η Επιτροπή ενέκριν, ε, ε, εντολή, διαπραγματευτική εντολή για το άνοιγμα συζητήσεων και διαπραγματεύσεων με την Τουρκία σε σχέση με τον εξυγχρονισμό της Τελειονικής Ένωσης και τη διεύρυνση των εμπορικών σχέσεων μεταξύ Ένωσης και Τουρκίας. Η συζήτησή μας σήμερα έχει ως ε, στόχο την ε, σύνταξη κατευθυντηρίων γραμμών, συστάσεων μάλλον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη διαπραγμάτευση. Και με αυτά θα ήθελα να δώσω το λόγο στον εισηγητή μας, τον κύριο Μπορέλη. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πριν περάσω στην ουσία του συζήτηση, θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι το πλαίσιο στο οποίο ε, συζητούμε εγγράφεται στο έγγραφο εργασίας ε, που ε, υλοποίησαμε τον Νοέμβριο και τα ουσιαστικά στοιχεία συνοψίζονται ως εξής. Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης ξεκινά από το γενικότερο θεματολόγιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στόχος θα πρέπει να είναι να ε, προωθεί τι αξίες και τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εμπορική πολιτική το ε, προσπαθεί να το επιτύχει αυτό μέσω συγκεκριμένων στόχων και μέσων τη εντολή τους. Η δράση της Επιτροπής εντάσσεται στο πλαίσιο της γενικότερη στρατηγικής ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να καθορίσουμε τι συγκεκριμένε πτυχέ, Δεν μπορούμε να παραβλέψουμε την συνολική κατάσταση της Τουρκία σήμερα. Το έγγραφο το οποίο θα αναλύσουμε σήμερα θέλει να εφαρμόσει στην πράξη αυτές τις υποδείξεις. Όπως είδατε, έχουμε διαρθρώσει σε τρεις ενότητες, οι οποίες είναι συντονισμένες μεταξύ τους και προχωρούν βαθμιδών. Πρώτα βλέπουμε τη γενικότερη κατάσταση και το πεδίο εφαρμογή. Στο δεύτερο σημείο έχουμε την ε, τελωνιακή εναρμόνιση και στο τρίτο μέρος ε, ε, εστιαζόμαστε στο εμπορικό σκέλος. Υπάρχει και μια τελική ενότητα που βλέπουμε τους στόχους αυτής της απόφασης. Όσον αφορά το γενικότερο πλαίσιο και το πεδίο εφαρμογή, ε, θελήσαμε να επισημάνουμε ότι η Τουρκία είναι στρατηγικό εταίρο τη Ευρωπαϊκή Ένωση, μεν, αλλά η ενίσχυση των εμπορικών σχέσεων θα πρέπει να γίνει βάσει κοινή βούληση να υπενθυμίσουμε τι αρχέ και τι ε, αξίε των συνθήκων τη Ευρωπαϊκή Ένωση οι διαπραγματεύσεις, παρά το γεγονός ότι στόχο έχουν ε, ένα ε, μελλοντικό πλαίσιο, γίνονται σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή και πρέπει να ληφθεί υπόψη η πολιτική, θεσμική και κοινωνική κατάσταση της Τουρκίας και να ζητήσουμε προστασία των αξιών και των Ευρωπαίων παραγωγών. Η συμφωνία στην οποία θα καταλήξουμε θα πρέπει να είναι πλήρης και άμεση και να ε, ε, ξεπεράσουμε καταστάσεις τις οποίες ε, ε, επιβάλαμε μονομερό στην Κύπρο. Επίσης, η δομή της Άγκυρας αυτή τη στιγμή είναι ακατάλληλη για το σημερινό πλαίσιο και την έχουν ξεπεράσει οι εμπορικές πολιτικές. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να συμμετέχει ενεργά και να παρακολουθεί και να αξιολογεί τις ε, συνέπειες των διαπραγματεύσεων και στην Τουρκία και στην Ευρώπη. Αυτό θα δώσει μεγαλύτερη νομιμοποίηση στην ίδια της διαδικασία της διαπραγμάτευσης και θα επιτρέψει να καθορίσουμε ένα διάλογο ο οποίος δεν υπήρχε υπήρξε στο ε, πρόσφατο παρελθόν μεταξύ τουρκική κυβέρνηση και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η Τελωνιακή Ένωση για να υλοποιηθεί θα πρέπει να σταματήσουν από πλευρά Τουρκία ε, ε, τα προστατευτικά μέτρα τα οποία εφάρμοσαν τα τελευταία χρόνια, να υπάρξει πραγματική ευθυγράμμιση με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και καταπολέμηση τη παραπία και, και του λαθρεμπορίου. Και επίση θα πρέπει να βρούμε έναν κατάλληλο μηχανισμό επίλυση διαφορών και να βελτιώσουμε τη συνεργασία στην ε, διαδικασία λήψη αποφάσεων κοινού συμφέροντο. Όσον αφορά τα πρόσφατα γεγονότα, θέλαμε να υπενθυμίσουμε για το εμπόριο ότι η απελευθέρωση των υπηρεσιών και των ε, κρατικών προμηθειών σημαίνει ότι οι τουρκικέ αρχέ θα πρέπει να ανοίξουν πλήρω τον ανταγωνισμό. Η απελευθέρωση θα πρέπει να γίνει σταδιακά και με δεσμευτικό τρόπο και να λάβουμε υπόψη και τι συνέπειε για τι μικρομεσαίε επιχειρήσει, του εργαζομένου, του καταναλωτέ και το περιβάλλον θα πρέπει να υπάρξει μια πραγματική εναρμόνιση στον τομέα ε, φυτογειονομίας και γεωργίας και επίσης ε, να ε, προστατεύσουμε κυρίως τα γεωργικά προϊόντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι ανοιχτά στον ανταγωνισμό. Θα πρέπει να γίνουν με σαφή κριτήρια διαφάνειας, αμοιβαιότητας και βάση των κριτηρίων του θετικού καταλόγου. Να αποκλειστούν οι οπτικοακουστικές υπηρεσίες και αυτές του γενικού οικονομικού συμφέροντος και επίσης να προσέξουμε την προστασία των δεδομένων και των επενδύσεων. Θα πρέπει να εγγυηθούμε τις διαδικασίες για την ε, είσοδο και παραμονή των επαγγελματιών και επίσης θα πρέπει ε, να γίνεται ε, σε συνθήκες ε, ανταγωνισμού ε, διαφάνειας. Επίσης, πέραν των τεχνικών στοιχείων, η έκθεση αυτή θέλει να διαβιβάσει προς το Συμβούλιο ότι το Κοινοβούλιο, παρά το γεγονός ότι θεωρεί ότι η διαδικασία προσχώρησης έχει παγώσει, θεωρεί ότι είναι στρατηγική σημασία να γίνεται διάλογος με την Τουρκία. Ο διάλογος για τον εμπορικό τομέα είναι χρήσιμος, δυνατόν να υλοποιηθεί και έχει και μεγάλη ουσία, αλλά θα πρέπει να συνεισφέρει σε ευρύτερε και συνολικότερε καταστάσεις. Θα πρέπει η διαπραγμάτευση να γίνεται ε, δεχόμενη το εξή, ε, γνωρίζοντας ότι θα υπάρχουν συνέπειες στο μέλλον. Και ε, αυτό το οποίο περιμένουμε είναι ένα νομοθετικό πλαίσιο το οποίο να είναι πραγματικά πιο ανταγωνιστικό, πιο ε, διάφανο και ε, θα πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένα μετρήσιμα μεγέθη για τους πολίτες, τους εργαζομένους και το περιβάλλον και τέλος ότι ο στόχος της διαπραγμάτευσης είναι μια θετική συμφωνία την οποία θα συμμερίζονται και οι δύο πλευρές αλλά δεν είναι δεδομένη αυτή η διαπραγμάτευση και μπορεί να υπάρξουν και άλλες δυνατότητες συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Τουρκίας. Τέλος, θέλουμε να διευκρινίσουμε όλο αυτό στο τελευταίο τμήμα και θεωρούμε ότι πρέπει ε, να δούμε λίγο και το χρονοδιάγραμμα αυτής της διαδικασίας. Η Γραμματεία με ενημέρωσε ότι κάποιες ε, πολιτικές ομάδες θα ήθελαν να αναβάλουν την ψηφοφορία στην Επιτροπή και στην Ολομέλεια με το επιχείρημα ότι οι αποφάσει μα για το θέμα αυτό δεν μπορούν να ε, χρησιμοποιηθούν με την ευκαιρία του δημοψηφίσματο που θα γίνει στην Τουρκία ε, σύντομα. Αυτό βέβαια ναι μεν είναι θεμητό, αλλά και το Συμβούλιο θα πρέπει να εγκρίνει την εντολή του πριν από την τελική μας ψηφοφορία, εάν τελικά αναβάλουμε εμείς την ψηφοφορία. Ως εισηγητής λοιπόν θα ήθελα να επισημανώ ότι πρώτο μας μέλημα θα πρέπει να είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ακουστεί στο συγκεκριμένο θέμα. Και επομένω, παρά το γεγονό ότι αντιλαμβάνομαι τα επιχειρήματα αυτών που ζητούν αναβολή, κατά την άποψή μου είναι να τηρήσουμε το χρονοδιάγραμμα, γιατί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να ε, πει και αυτό την άποψή του εγκαίρως. Θα μπορούσαμε ίσως να αλλάξουμε αν υπάρξει συγκεκριμένη δέσμευση του Συμβουλίου να περιμένει την άποψη του Κοινοβουλίου. Ε, επειδή δεν υπάρχει τέτοια βεβαιότητα αυτή τη στιγμή, δεν μπορούμε να εκθέσουμε το Κοινοβούλιο στον κίνδυνο να μην ακουστεί άποψή του σε ένα τόσο σημαντικό θέμα και όχι μόνο για τα εμπορικά θέματα. Γι' αυτό ακριβώ και ζητώ να διατηρήσουμε το χρονοδιάγραμμα. Τώρα, εάν κάποιο θέλει να χρησιμοποιήσει τι αποφάσει μα με κατάλληλο τρόπο, θα φροντίσουμε να εξηγήσουμε για ποιο λόγο έγινε η δουλειά μα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ο λόγος τώρα στους Σκιώδης. Πρώτα από το ΕΛΚ. Ο Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Μπορέλη για τις εκτενείς και ε, του, για την εκτενή του προσέγγιση, για την, τον επαγγελματισμό με τον οποίο προσεγγίζει το θέμα της Τελειονικής Ένωσης με την Τουρκία. Δεύτερον, νομίζω ότι είναι σαφές σε όλους μας, εδώ στο Κοινοβούλιο αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση ευρύτερα, ότι η Τουρκία αυτή τη στιγμή ε, διέρχεται μια τεράστια πολιτική αλλά και οικονομική ε, διαδικασία αλλαγών. Θεωρώ ότι πρέπει να ε, ότι οι δυνατότητες μας να προωθήσουμε τα δικά μας θέματα στην Τουρκία αυτή τη στιγμή είναι περιορισμένες. Για λόγους που δεν χρειάζεται να αναφέρω και να αναλύσω εδώ. Σε κάθε περίπτωση ο εξυγχρονισμός της Ελληνικής Ένωσης είναι σημαντικός να γίνει διότι μπορεί να λύσει και να βελτιώσει την ε, κατάσταση ε, όσον αφορά τις εμπορικές και οικονομικές μας σχέσεις, αλλά ταυτόχρονα μπορεί να αυξήσει, αν δράσουμε με σοφία, την επιρροή μας στα όσα συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στην Τουρκία. Και αυτό δεν είναι μικρό ζήτημα. Αν λάβει κανείς υπόψη του το επικείμενο δημοψήφισμα, τις ε, διαπραγματεύσεις για την ε, ιστορική επανένωση της Κύπρου κτλ. κτλ. Από αυτή την άποψη λοιπόν, διαβάζοντας το σχέδιο έκθεσης που ε, μας παρουσίασε με εξαιρετικό τρόπο ο κύριος Μπορέλη, έχω κάποιες μικρές αλλά σημαντικές θα έλεγα προσθήκες, τις οποίες και προτείνουμε ως Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και αυτές είναι 5-6 αλλαγές στην ουσία. Χρειαζόμαστε νομίζω κάποιες βελτιώσεις και κάποιες προσθήκες όσον αφορά τις δεσμεύσεις της Τουρκίας για να αποδείξει την προθυμία της να προχωρήσουμε μπροστά. Επίσης ε, υπάρχει μια προσθήκη που αφορά την εφαρμογή των ήδη συμφωνηθέντων μεταξύ Ένωσης και Τουρκίας ε, στους τομείς που ενδεχομένως υπάρχουν κάποιες αμφιβολίες ή και κάποια πισωγυρίσματα. Ε, ειδικό κεφάλαιο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που πιστεύουμε ότι θα πρέπει να υπάρχει. Σημαντικό θέμα είναι και οι κανόνες διαφάνισης για τους ε, ε τομείς με υψηλό βαθμό ρύθμισης μέτρα ε, για την υγεία των ανθρώπων και των φυτών και τέλος γενική πολιτική διάσταση του εξυγχρονισμού της Τελωνιακής Ένωσης. Αν λάβουμε υπόψη μας όλα αυτά τα θέματα, πιστεύω ότι μπορούμε να προχωρήσουμε ε, και να επιτύχουμε τον εξυγχρονισμό της ε, Τελωνιακής αυτής Ένωσης με την Τουρκία. Τουλάχιστον αυτό είναι πρόταση της δικής μου ομάδας. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα εκ μέρους των σοσιαλιστών, Γιος Ντάντι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τον συνάδελφο Βορέλη για την δουλειά του και ε, να πω ότι εγώ θεωρώ ότι η έκθεση αυτή αποτελεί πολύ καλή βάση και όσον αφορά τον πιθανό εξοχρονισμό της Τελωνιακής Ένωσης, αλλά και την επέκταση των εμπορικών σχέσεων μεταξύ ε, ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκία, ε, γιατί θα ανοίξουν κεφάλαια που αφορούν τη γεωργία, τις υπηρεσίες, τις κρατικές προμήθειες. Εμείς θα υποβάλουμε κάποιες τροπολογίες για να ενισχύσουμε κάποια τμήματα. Θα επανέλθω σε αυτό αργότερα βέβαια, γιατί θα ήθελα να ξεκινήσω με το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή, όπως υπενθύμησαν αρκετοί στις παρεμβάσεις τους, δεν είναι κατάλληλη στιγμή και δεν υπάρχει κατάλληλη χρονική συγκυρία αυτή τη στιγμή γιατί είναι ευαίσθητε οι σχέσει μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας. Όσον αφορά το ε, την απόπειρα πραξικοπήματο. υπήρξαν συγκεκριμένε παραβιάσει ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη συνέχεια και ελευθεριών στην Τουρκία και μετά μια σταδιακή επιδείνωση της κατάσταση του κράτους δικαίου και αυτό φυσικά ε, έρχεται να κορυφωθεί με το δημοψήφισμα που θα γίνει στα, ως, ε, στην Τουρκία στη συνέχεια. Οι συνθήκε λοιπόν δεν είναι καθόλου ευνοϊκέ. Η στρατηγική του εισηγητή να εκφράσει την άποψή του το Κοινοβούλιο πριν δοθεί η διαπραγματευτική εντολή από το Συμβούλιο. Ε, με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο. Άκουσα αυτά που είπε ο Συγητή ε, για το χρονοδιάγραμμα και εγώ πιστεύω ότι το χρονοδιάγραμμα θα πρέπει υποχρεωτικά ε, με πιέσεις και προς το Συμβούλιο να ε, πάρει μια αναβολή ώστε να μπορέσει και το Κοινοβούλιο να κάνει αυτό που το αναλογεί για να εκφράσει την άποψή του ε, πριν το Συμβούλιο ε, δώσει διαπραγματευτική εντολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά ταυτόχρονα δεν θα πρέπει να επηρεάσει και τις εσωτερικές πολιτικές δυναμικές ε, της Τουρκίας ε, και ιδιαίτερα το δημοψήφισμα. Γι' αυτό λοιπόν και ελπίζω το Συμβούλιο να δώσει ε, κάποια ένδειξη ότι είναι διατεθειμένο να βοηθήσει και προς αυτή την κατεύθυνση το Κοινοβούλιο. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι η Τουρκία είναι υποψήφια χώρα από το 2005 και περιμένουμε με ακόμα μεγαλύτερο σθένος προστασία δικαιωμάτων που αποτελούν και τη βάση της Ένωσής μας. Η εμπορική πολιτική μας θα πρέπει να είναι συνεπής με το σύστημα των αξιών που μας χαρακτηρίζει και θα πρέπει αυτό να το αποδεικνύουμε ε, πάντα, αλλά κυρίως σε αυτή την περίπτωση. Και τώρα θα ήθελα να περάσω στην ουσία και να κάνω κάποιε σκέψει. Καταρχά, η Τελωνιακή Ένωση υπάρχει, αλλά δεν λειτουργεί σωστά. Ε, και επομένως, ε, ο εξυγχρονισμό σημαίνει ωφέλη και για τι δύο πλευρές, ιδίως ε, αν καταφέρουμε να έχουμε όλο και μεγαλύτερη ευθυγράμμιση τη Τουρκία με το κοινωνικό κεκτημένο και επομένω να έχουμε και μεγαλύτερη ολοκλήρωση. Παρά το γεγονό ότι είχαμε κάποιε πρόσφατε εξελίξει, οι εμπορικέ σχέσει μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Τουρκία θα συνεχίσουν να υπάρχουν ε, και ε, το νομικό σύστημα ε, όμως είναι παροχημένο αυτή τη στιγμή. Η Τελωνιακή Ένωση είναι τελείως διαφορετική πραγματικότητα και παράλληλη με τη διαδικασία ένταξης. Το Νοέμβριο ζητήσαμε να παγώσει η διαδικασία διαπραγμάτευσης με την Τουρκία και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει ένας ανοιχτός διάβλος επικοινωνίας και αυτό είναι σίγουρα ένα πολύ σημαντικός ε, διάβλος. Δεν μπορούμε να αποφασίσουμε να κόψουμε τελείως γέφυρες με μια χώρα με την οποία έχουμε ε, συνάψει συμφωνία για τη μετανάστευση πριν από κάποιου μήνε. και πρέπει να επενθυμίσω ότι δεν τους δώσαμε και ψυχία, του δώσαμε πάρα πολλού πόρου ε, για τη μετανάστευση και τη συμφωνία αυτή και επομένω πιστεύω ότι και από γεωπολιτική σκοπιά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μα αυτή την πτυχή και την προσέγγιση που υπήρξε αυτή την τελευταία περίοδο ε, της Τουρκίας με τη Ρωσία. Επίσης, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τον εξυγχρονισμό της Τελωνιακή Ένωση ως ένα εργαλείο στη διάθεσή μας για να ξεκινήσει μια ε, πορεία σταθερότητας, δημοκρατίας και ελευθερίας και προσέγγιση. Τη Τουρκία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μαζί με άλλους συναδέλφους λοιπόν θα σας υποβάλω μια σειρά από τροπολογίε, οι οποίες επικεντρώνονται σε κάποια σημεία. Πρώτον, ο εξυγχρονισμό της Τελωνιακή Ένωσης και η επέκταση των εμπορικών σχέσεων που θα μπορούσαν να αποτελέσουν πολύ σημαντικό διάβλο για να μετριάσουμε τι πολιτικέ εντάσει και να υπάρξει και ε, προστασία για να μην υπάρξει επιδείνωση των σχέσεων με την Τουρκία. Πρέπει να επιλύσουμε ό,τι δεν λειτουργεί, ξεκινώντα από ένα αποτελεσματικό μηχανισμό επίλυση διαφορών και να εμβαθύνουμε τι εμπορικέ σχέσει με την κατάλληλη προστασία των πιο ευαίσθητων τομέων. Ζητάμε από την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει στι διαπραγματεύσει όλα τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μα προκειμένου να επηρεάσουμε όσο μπορούμε την Τουρκία σε θέματα προστασία ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κυρίω σε θέματα προστασίας των δικαιωμάτων των πολιτών και των εργαζομένων, όπως για παράδειγμα την προσθήκη μιας ρήτρας αναστολής που αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες και ένα κεφάλαιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη που περιλαμβάνει δεσμευτικέ διατάξεις και ένα μηχανισμό κυρώσεων. Τέλος, Κάτι πάρα πολύ σημαντικό για τη ε, σύναψη της συμφωνίας θα πρέπει να είναι η πλήρη εφαρμογή για όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με πρώτο και καλύτερο την Κύπρο. Ολοκληρώνοντας πιστεύω ότι η μεγάλη αξία αυτής της έκθεσης ε, έγκυται ακριβώς στο γεγονός ότι το Κοινοβούλιο μπορεί να εκφράσει σαφή θέση για την έναρξη αυτών των διαπραγματεύσεων και ελπίζουμε ότι ε, θα μπορέσουν να αντανακλούν και τις δικές μας τις θέσεις. Ευχαριστώ τους συναδέλφους για τη συνεισφορά τους και ελπίζω να μπορέσουμε να έχουμε επικοδομητική συνεργασία στις τροπολογίες. Thank you very much and I turn now to... Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ε, θα μιλήσω εκ μέρους ε, του καθηγητή Στάρβατη τα σχόλιά του ουσιαστικά είναι ερωτήσει ε, που δείτε προ την Επιτροπή, οπότε ελπίζω πω θα μπορέσει να μα απαντήσει. Η Τουρκία λοιπόν έχει εκφράσει επανειλημμένα τι ανησυχίε τη για το γεγονό ότι, ότι ε, παρότι δεν συμμετέχει σε καμία ε, από τι συμφωνίε λήψη αποφάσεων τη Ευρωπαϊκή Ένωση, παρόλα αυτά καλείται να εφαρμόσει όλου του όλους τους κανόνες που ισχύουν σε ό,τι αφορά την Τελωνιακή Ένωση. Και πολλέ φορέ οι τρίτε χώρε αποθαρρύνονται από το να έρθουν σε διμερή διαπραγμάτευση με την Τουρκία γιατί απευθύνονται στην Επιτροπή για να εξασφαλίσουν ε, πρόσβαση στην ενιαία αγορά. Άρα λοιπόν η ε, Ποιο θεωρεί η Επιτροπή πω είναι ο κατάλληλο ε, τρόπο για να εμπλακεί σε αυτή τη διαδικασία η Τουρκία, αφού δεν αποτελεί πλήρε μέρο τη Ευρωπαϊκή Ένωση, πώ δηλαδή μπορεί να συμμετάσχει η σχετική χάραξη τη πολιτική, πώ μπορεί δηλαδή να ανταποκριθεί στι επιθυμίε αυτή τη Τουρκία. Και δεύτερο, σε ό,τι αφορά την επίλυση διαφορών, η Επιτροπή μπορεί να μα επιβεβαιώσει ότι θα βασιστεί στα υφιστάμενα μοντέλα ε, που ισχύουν στις σχετικές συμφωνίες για την επίλυση διαφορών, δηλαδή της ε, ελεύθερης, ε, του ελεύθερου εμπολίου και θα εφαρμόσει κάτι τέτοιο, για παράδειγμα σε σχέση με την Ουκρανία, για παράδειγμα συμφωνία που υπάρχει και όπου σχετικές αποφάσεις του δικαστηρίου θεωρούνται δεσμευτικές. Πώς θα επιτύχει μια τέτοια σύγκληση με την Τουρκία και πραγματικά ελπίζουμε να λάβουμε απαντήσεις από την Επιτροπή. Μαρή Κεσάκια για την άλλη έχετε το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ τον εισηγητή και ευχαριστώ και όλους τους προηγούμενους ομιλητές που με κάλυψαν σε μεγάλο βαθμό, οπότε θα είμαι σύντομη. Ε, νομίζω πως όλοι γνωρίζουμε καλά πόσο δύσκολη είναι η κατάσταση, ε, την οποία αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι στην Τουρκία μετά δηλαδή και από το αποτυχημένο πραξικόπημα ε, και μετά όσα προβλήματα υπάρχουν σε επίπεδο σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Άρα λοιπόν το Κοινοβούλιο θα πρέπει να συνεχίσει να ασχολείται με αυτά τα ζητήματα. Από την άλλη πλευρά θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι πραγματικά ε, το γεγονός ότι Τελωνιακή Ένωση είναι πλέον παροχημένη ε, και αυτό επηρεάζει και εμά εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα λοιπόν είναι σημαντικό να συνεχίσουμε τι προσπάθειέ μα για εξυγχρονισμό ε, του ε, Τελωνιακού Κώδικα προκειμένου να παρέχουμε καλύτερε υπηρεσίε και οι σχετικοί κανόνε να ανταποκρίνονται στην σύγχρονη οικονομία στην οποία ζούμε σήμερα. Επίση θα πρότεινα να αξιοποιήσουμε αυτή τη διαδικασία έτσι ώστε να έρθουμε επικοδομητικά, δημιουργικά σε επαφή με την Τουρκία, αφού δεν μα δίνονται πολλέ τέτοιε ευκαιρίε. Δηλαδή, αναφέρθηκε η Συμφωνία για το Μεταναστευτικό, ε, ε, για την οποία εγώ υιοθετώ επικριτική στάση, αλλά παρόλα αυτά ω ε, γειτονικέ περιοχέ, γειτονικέ χώρε έχουμε πολλού τέτοιου δεσμού πολιτισμικού, οικονομικού και πολιτικού και κατά συνέπεια θα πρέπει να αξιοποιούμε τέτοιε ευκαιρίε για να βρισκόμαστε σε επαφή με αυτή τη γειτονική χώρα. Ε, συμφωνώ σε γενικές γραμμές με τα όσα μας προσφύγει και ειδικότερα ε, την έκκληση που εξέφρασε να μην καθυστερήσουμε περαιτέρω τη σχετική διαδικασία. Δηλαδή υπάρχει ο κίνδυνος να υπάρξουν επιμέρους μικροκαθυστερήσεις ενώ ε, Εκείνο που θα έπρεπε αντιθέτω να κάνουμε είναι να χρησιμοποιήσουμε το ενδιαφέρον που υπάρχει για να επιτύχουμε αυτόν τον εξυγχρονισμό τη Τελωνιακή Ένωση. Υποστηρίζω λοιπόν την προσέγγιση του εισηγητή ε, και βέβαια υπονθυμίζω πως η έναρξη των διαπραγματεύσεων είναι ένα πράγμα, το κλείσιμο, η οριστικοποίηση των διαπραγματεύσεων είναι άλλο πράγμα. Οπότε ας ξεκινήσουμε αυτή τη διεργασία που πρέπει να ξεκινήσουμε και θα δούμε από εκεί και μετά πού θα μας πάει. Ε, ο κύριος Ερσόλτς έχει τώρα το λόγο εκ μέρους της ΓΚΟΕ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, θα μιλήσω εκ μέρου ε, του κ. Στέλιου Κούλογλου, που είναι ο σκιώδη ε, της τη ομάδα μα, ο οποίο δεν κατέφερε να παρευρεθεί σήμερα εδώ και γι' αυτό θα διαβάσω τη δική του παρέμβαση. Όμω, προτού το κάνω, θα ήθελα να ρωτήσω λίγο τον κύριο Μπορέλ και βασικά σε σχέση με το σχόλιο που έκανε σε ό,τι αφορά την καθυστέρηση ή όχι τη δική μα τοποθέτηση. Αντιλαμβάνομαι την πρόταση που έκανε η σοσιαλιστική ομάδα, αλλά Εάν θέλουμε το Κοινοβούλιο να επηρεάσει την θέση της Ένωσης σε σχέση με αυτό το ζήτημα θα πρέπει να το κάνει πρωτού υπάρξει μια συμφωνία. Άρα δηλαδή υπάρχει ένα συγκεκριμένο χρονικό ε, περιθώριο το οποίο θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας. Οπότε το, το αναφέρω αυτό στον εισηγητή για να το λάβει υπόψη. Ο κύριο Σεκούλογλου λοιπόν λέει ότι κυρίε και κύριοι συνάδελφοι, να ευχαριστήσω ε, τον εισηγητή κύριο Μπορέλη για όλη την προσπάθεια που κάνει και όλε τι ιδέε που έχει συμπεριλάβει ε, σε αυτή την ε, πρόταση ψηφίσματο. Ωστόσο, υπάρχουν μία σειρά αποζητήματα τα οποία θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μα αν θέλουμε να προχωρήσουμε σε μία εξυγχρονισμένη τελωνιακή ένωση μεταξύ Ένωση και Τουρκία. Καταρχήν, θα πρέπει να ευθυγραμμιστεί σε επίπεδο νομοθεσία με το κεκτημένο, το κοινοτικό κεκτημένο σε σχέση με την ενωσιακή νομοθεσία και θα πρέπει προφανώς η Τουρκία καταρχήν να αντιποκριθεί στις διμερείς υποχρεώσεις που έχει αναλάβει και να σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα προτού ε, περάσουμε ε, σε περαιτέρω συμφωνίες. Επίσης ε, θα πρέπει να απελευθερώσει όλα τα κρατούμενα μέλη του, ε, του πολιτικού κόμματος της και ειδικότερα του Πρόεδρου. Επίσης ε, προτού ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις ε, με την ε, Τουρκία να διευκρινιστούν αυτά τα ζητήματα και γι' αυτό ε, ε, ζητώ πρωτού ξεκινήσει η σχετική επίσημη διαπραγμάτευση με την Τουρκία να διευκανθούν αυτά τα θέματα. Ε, εκ μέρου λοιπόν τη NGO NGL δεν υποστηρίζουμε την Τελωνική Ένωση ό,τι αφορά την, και την απέλευση ό,τι αφορά τις μεταφορέ, την αυσιπλοεία, τις δημόσιε προημήθειε και άλλου τομεί. Επίση, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μα ότι εξωτερικές, ή μάλλον, εξωτερικέ σχέσει και η εμπορική πολιτική όπω αναφέρθηκε και από από άλλους συναδελφούς σήμερα, θα πρέπει να συμβάλλουν ε, στην βιώσιμη ανάπτυξη, στην εξάλληψη της φτώχειας, στην προώθηση της δημοκρατίας, το κράτος δικαίου και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ε, πράγμα το οποίο αποτελεί και στρατηγική την οποία έχει ασπαστεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Άρα λοιπόν το θέμα που συζητούμε σήμερα της Τελωνιακής Ένωσης ε, με την Τουρκία δεν έχει να κάνει μόνο με εμπορικές πτυχές αλλά και με πολιτικές τεχνικού χαρακτήρα θέματα. Οπότε θα ήθελα να ζητήσω από την Επιτροπή και το Συμβουλίο να μην ξεκινήσει κάποια διαπραγμάτευση σε ό,τι αφορά την και Ένωση μέχρι ότου να διασφαλίσει το σεβασμό του κράτου δικαίου ε, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τη Δημοκρατία ή Τουρκία από την πλευρά τη. Ευχαριστώ και η απελευθέρωση ενδεχομένω του Τούρκου και Γερμανού ε, δημοσιογράφου την πλευρά τη Τουρκία θα μπορούσε να αποτελέσει μια πάρα πολύ ε, καλή πρώτη κίνηση. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Ε, η ομάδα μου πιστεύει ότι είναι απαραίτητο να εξευρεθούν τρόποι για να επηρεάσουμε την δραματική κατάσταση και την έλλειψη κράτους δικαίου ε, καθώς και της λειτουργίας της κοινωνίας των πολιτών στην Τουρκία ώστε η χώρα αυτή να πιστεί ότι είναι ανάγκη να επιστρέψει στον δημοκρατικό δρόμο και να αποφασίσει να επαναπροσεγγίσει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρ' όλα αυτά, πιστεύουμε ότι η κατάσταση έχει διαμορφωθεί με τέτοιον τρόπο, ώστε ο πρόεδρος Ερντογάν δεν ενδιαφέρεται ιδιαίτερος για τα όσα έχει να πει σε αυτά τα θέματα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ενδεχομένω, ο εξυγχρονισμός Ένωση Ένωσης ε, θα, ε, πρέπει, ε, θα μπορούσε ενδεχομένως να είναι το μοναδικό μας εργαλείο προκειμένου να δείξουμε την δυσαρέσκειά μας για τι εξελίξεις στην Τουρκία καθώς ο Ερντογάν προφανώς έχει αποδείξει ότι δεν ενδιαφέρεται για τις απόψεις μας σχετικά με την δημοκρατία, το κράτος δικαίου, το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα του. Πιστεύω επίσης ότι ε, καθώς υπάρχουν ε, ε, ε, κάποιες ε, σκέψεις για αναβολή της ψηφοφορίας, ε, να, ότι θα ήταν καλό να υπάρξει αναβολή και της προθεσμής υποβολής τροπολογιών. Ευχαριστώ πολύ από το ΙΕΝΕΦ. E Δυστυχώς ε, πρέπει να ομολογήσω ότι δεν παρακολούθησα ε, ε, μάλλον παρακολούθησα με προσοχή τη συζήτηση και μου φαίνεται περίεργο αυτό που συμβαίνει εδώ γιατί ο καθένας προσπαθεί από ό,τι μου φαίνεται να χαράξει ένα δρόμο ισορροπίας ε, και ε, μάλιστα είναι πολύ πρόθυμοι να θυσιάσουν την δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα στο βωμό ε, των εμπορικών σχέσεων με την Τουρκία. Μια στάση η οποία δεν, την οποία δεν επέδειξαν πολύ στη Ρωσία, η οποία είναι πολύ σημαντικότερος εμπορικός εταίρος. Εκεί εξάντλησαν την αυστηρότητά τους μερικοί, ε, και αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι σε αυτή την περίπτωση η Τουρκία πραγματικά μόνο κερδισμένη μπορεί να βγει από έναν τέτοιον εξορονισμό της Τελωνιακή Ένωσης. Γνωρίζετε ότι ε, ε, η Τελωνιακή Ένωση αυτή και ο εξεχρονισμός της θα ε, στρώσουν το έδαφος για την είσοδο διαφόρων απορροκυπευτικών της Τουρκίας στην ευρωπαϊκή αγορά. Το ίδιο και σχέση σε σχέση με τα παραποιημένα προϊόντα, με τι απομιμήσει. Ε, για μένα η Τουρκία δεν είναι ευρωπαϊκό κράτος ε, και γι' αυτό δεν υπάρχει και πιο, ε, κανένας λόγος να τις επιτρέψουμε να μπει από το πίσω παράθυρο ε, μέσω της ε, Τελωνιακής Ένωσης. Νομίζω ότι κάτι τέτοιο θα ήταν πάρα πολύ άδικο και δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να το επιτρέψουμε. Ευχαριστώ λέει ο Πρόεδρος και τώρα ο λόγος στα μέλη της Επιτροπής μας. Παρακαλώ. Συνάδελφοι. Εκτός μικροφώνου η ομιλήτρια. Ωραία. Ε, αυτή τη στιγμή η Τελωνιακή Ένωση γνωρίζουμε ότι δεν λειτουργεί ούτε τεχνικά ούτε πολιτικά. Το γνωρίζουμε αυτό. Η κατάσταση είναι ε, πράγματι δύσκολη στην ε, Τουρκία. Εμείς ωστόσο ε, ε, υποστηρίζουμε την Τελωνιακή Ένωση. Αλλά το τονίζω, εξυγχρονισμός της Τελωνιακής Ένωσης, όχι η Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου. Για μας τρία σημεία είναι σημαντικά. Πρώτον, διαφάνεια, δηλαδή θα πρέπει η εξυγχρονισμένη έκδοση τη Ελληνική Ένωση να δημοσιευθεί αμέσως μετά την ε, υπογραφή της και θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα, οι απόψεις του Κοινοβουλίου. Ε, για την απελευθέρωση των, ε, ε της παροχής υπηρεσιών θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να εξαιρεθούν οι, οι μεταφορές. Ε, όσον αφορά το, τον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των εργασιακών δικαιωμάτων είναι ένα ζήτημα που πραγματικά πρέπει οπωσδήποτε να κατοχυρωθεί μέσα στη συμφωνία ενώ αν υπάρξουν παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή περιορισμός της ε, ελευθερίας της έκφρασης θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα προσωρινής έστω αναστολής της συμφωνίας. Και ε, σε περίπτωση που γίνουν τέτοια πράγματα κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων θα πρέπει οι διαπραγματεύσεις να παγώσουν. Γενικά ε, θεωρούμε ότι αυτά τα κριτήρια θα πρέπει να προσδιοριστούν πριν από την, ε, πριν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων ιδίω όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ε, ε, επίσης απορρίπτουμε αυτό το καθεστώς παρατηρητή ε, που πρόκειται να αποδοθεί στην Τουρκία. Ο κύριος Μαυρίδης έχει το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν θέλω να δώσω τα συγχαρητήρια μου στον συνάδελφο τον κύριο Ντέιβιτ Πορέλη για την προσπάθεια που κάνει να συγκεράσει διαφορετικές απόψεις σε ένα πολύ δύσκολο θέμα, ομολογουμένως. Ε, όποτε μιλάμε, κύριε Πρόεδρε και κύριοι συνάδελφοι, για την Τελωνιακή Ένωση της Τουρκίας, είναι μια πονεμένη ιστορία. Είναι μια ιστορία με πολλά προβλήματα. Και θα είμαι πάρα πολύ σύντομος, αλλά θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω λέγοντας ότι υπάρχει ήδη μια υφιστάμενη αρχική συμφωνία τελωνιακής σύνδεσης Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας και η Τουρκία τότε δεσμεύτηκε ενώπιον όλων μας και των 28 κρατών μελών ότι θα εφαρμόσει τη συμφωνία εκείνη με όλα τα κράτη-μέλη χωρίς διακρίσεις. Και όμως την επομένη με δήλωσή της ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να την εφαρμόσει με την Κυπριακή Δημοκρατία. Ένα ισότιμο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και το ερώτημα είναι με ποιο εχέγγυο θα πρέπει να ξαναεμπιστευτούμε μια διαδικασία αναβάθμισης των εμπορικών σχέσεων με την Τουρκία και της αναβάθμισης της Ελληνική Ένωσης. Και αυτό με οδηγεί στο δεύτερο σημείο, που με βρίσκει σύμφωνο με κάτι που είπε ο συνάδελφός μου, ο Νικολάη Τάντι. Εμείς εδώ έχουμε εμπορικά συμφέροντα, αλλά το μέγιστο συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι the respect of the rule of law. Και διαρωτώ με, σε σχέση με μας ως Ευρωπαϊκή Ένωση, ποια είναι, ποιος είναι ο καλύτερος, το καλύτερο εχέγγυο, ποια είναι η καλύτερη εγγύηση ότι αυτή τη φορά η Τουρκία, εάν ξεκινήσουμε αυτή τη διαδικασία, θα εφαρμόσει τη συμφωνία. Νομίζω ότι η το καλύτερο εχέγγυο είναι ένα, να εφαρμόσει ήδη την υφιστάμενη συμφωνία και αυτό είμαι βέβαιος ότι θα απαιτούσε και ο κάθε συνάδελφος για το δικό του κράτος μέλος. Τελειώνω με μια κουβέντα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, επειδή ήδη λέχθηκε από πάρα πολλούς συναδέλφους και με βρίσκουν 100% σύμφωνοι. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, οι συνθήκες γύρω από τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Τουρκία ολοένα και χειροτερεύουν. Το καθεστώς Ερτογάν, φυσικά όπως κάθε καθεστώς, προσπαθεί να εμπεδώσει την εξουσία του. Εμείς θα αναλάβουμε πρωτοβουλία για να προσφέρουμε αναβάθμιση στην οικονομία της, αυτού του καθεστώτος για να εμπεδώσει την εξουσία του ή θα κινηθούμε τουλάχιστον παραμένοντας παθητικοί. Τελειώνω με μια τελευταία παρατήρηση. Κοιτάζοντας το κείμενο, έχω αντιληφθεί ότι παρόλο που είναι γύρω από εμπορικές σχέσεις, υπάρχουν και νομικά και πολιτικά ζητήματα. Για παράδειγμα, η αναγνώριση της Κυπριακής Δημοκρατίας από την Τουρκία και η εφαρμογή της Τελωνιακής Ένωσης και με την Κυπριακή Δημοκρατία είναι νομική υποχρέωση. Δεν είναι θέμα πολιτικής άποψης. Και το δεύτερο είναι ότι πώς μπορούμε σε ένα τέτοιο κείμενο να προτείνουμε ή να εισηγούμαστε καθεστώς παρατηρητή στην Τουρκία στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέσα σε όλη αυτή τις συνθήκες που έχουμε περιγράψει. Νομίζω για μένα τα πράγματα είναι πεντακάθαρα. Τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αυτά που υπερέχουν καλά τα υπόλοιπα συμφέροντα, αλλά αν θέλουμε να έχουμε μέλλον πρέπει να ξεκινήσουμε με τον σεβασμό των βασικών κανόνων δικαίου. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Uh, thank uh, Σας ευχαριστώ πολύ. Υπάρχουν άλλα σχόλια. Όχι, να, να δώσουμε το λόγο στην Επιτροπή. Ο κύριος Γκαρθία Μπερθέντου. Ευχαριστώ πολύ και θα ήθελα να ξεκινήσω ευχαριστώντας τον εισηγητή και τα μέλη της Επιτροπής ε, για μια πάρα πολύ σημαντική έκθεση και για τα σχόλια τα οποία ακούσαμε. Θα ήθελα να σας ε, κάνω κάποια σχόλια σε σχέση με τα όσα ακούσαμε σήμερα το απόγευμα. Πρώτον, πρέπει να Είμαστε πολύ προσεκτικοί. Η Τουρκία είναι πολύ σημαντικό εμπορικό εταίρο. Είναι η τέταρτη μεγαλύτερη αγορά εξαγωγών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οι παρούσε εμπορικέ και οικονομικέ σχέσει είναι ασύμετρες ε, ε, προς το όφελος της Τουρκίας. Ε, ανοίξαμε την γεωργική μας ε, ρά ενώπιον της Τουρκίας ε, πολύ περισσότερο από ό,τι την έχουν αυτήσει ε, ενώπιον ημών. Υπάρχει μια ανοιχτή διαδικασία υποβολής ε, προσφορών σε μειοδοτικούς διαδικονισμού που δεν υπάρχει στην Τουρκία. Υπάρχουν πολλές υπηρεσίες στην Τουρκία οι οποίες δεν εφαρμόζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από μία άποψη λοιπόν πηγαίνουμε στην Ευρωπαϊκή, στις διαπραγματεύσεις αυτές με πολύ σημαντικά επιθετικά χαρτιά και θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι η Τουρκία θα ανοίξει πολύ περισσότερο ενώπιον της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με το τι κάνει αυτή τη στιγμή. Δεύτερον, θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι η Τελωνιακή Ένωση, ε, η οποία συμφωνήθηκε το 1995, είναι μια συμφωνία η οποία συνάφηκε πριν από πάρα πολύ καιρό και δεν ανταποκρίνεται αυτή τη στιγμή με την παρούσα προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το τι ακριβώς πρέπει να περιλαμβάνει μια σύγχρονη ε, προοδευτική εμπορική σχέση. Δεν υπάρχει καμία δέσμευση για τη βιώσιμη ανάπτυξη, δεν υπάρχει καμία δέσμευση στην Τελωνιακή Ένωση και στη Συμφωνία της Άγκυρας για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν έχουμε αυστηρούς κανόνες ε, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ε, για το SPS, ε, τη ρυθμιστική συνοχή και ο λόγος για τον οποίο οι διαπραγματεύσεις αυτές αποτελούν σημαντική ευκαιρία να εξυγχρονίσουμε τις εμπορικές μας σχέσεις με την Τουρκία και να είναι πολύ πιο κατάλληλη και βάσει των αξιών που προασπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και βεβαίως υπάρχει και το πρόβλημα ότι η Τελωνιακή Ένωση δεν λειτουργεί αποτελεσματική, μεταξύ άλλων γιατί δεν υπάρχει ένα ένας αποτελεσματικός μηχανισμός επίλυσης διαφορών. Μία από τις σημαντικές λοιπόν πτυχές που θέλουμε να καλύψουμε σε αυτές τις διαπραγματεύσεις είναι να έχουμε ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό μηχανισμό επίλυσης διαφορών και θα πρέπει να δούμε με ποιο τρόπο θα γίνει αυτό στι διαπραγματεύσει. Σημείωσε και τα ερωτήματα τη Emma Clarking όσον αφορά το μοντέλο με την Ουκρανία και είναι αλήθεια ότι αυτή τη στιγμή ε, πρέπει να λάβουμε υπόψη μα ε, θέματα αριθμιστικής ευθυγράμμαση, λαμβάνοντας υπόψη και το ρόλο του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Και το μοντέλο αυτό δεν ξέρω κατά πόσο θα πρέπει να το εξετάσουμε. Είναι λίγο νωρί αυτή τη στιγμή να δούμε ε, ε, τι μηχανισμό θα επιλέξουμε και πώς θα λειτουργεί. Επίσης είναι σαφές ότι θέλουμε σε αυτές τις διαπραγματεύσεις με την Τουρκία Εάν θέλουμε να πετύχουμε, θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να απαντήσουμε και στι ανησυχίε για το τι συμβαίνει με χώρε οι οποίε διαπραγματεύονται Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου με την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν διαπραγματεύονται με την Τουρκία. Θα πρέπει να βρούμε ε, μια ε, εφάνταστη απάντηση για να απαντήσουμε σε αυτή την ανησυχία της Τουρκίας, σεβόμενη όμως πλήρως την αυτονομία της εμπορικής πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Τουρκία δεν είναι κράτος μέλος και επομένω δεν μπορεί να διαδραματίζει τον ίδιο ρόλο με τα κράτη-μέλη για την ανάπτυξη της εμπορικής πολιτικής μας και ε, θα πρέπει να δούμε ακριβώς πώς θα χαράξουμε τη διαχωριστική γραμμή στις συζητήσεις και στις διαπραγματεύσεις. Βεβαίω συνειδητοποιούμε απολύτω και το πολιτικό πλαίσιο. Πιστεύουμε ότι η δέσμευση είναι πολύ καλύτερη στρατηγική από την ανυπαρξία δέσμευση, αλλά βεβαίως αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να υπερασπιστούμε στεναρά την Ευρωπαϊκή Ένωση και σε οικονομικού και σε πολιτικού όρου. και θα δείτε και ότι η εντολή που έχει ε, παρουσιάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρεται σαφέστατα στα ανθρώπινα δικαιώματα, αναφέρεται σαφέστατα στο βιώσιμη ανάπτυξη, αναφέρεται σαφέστατα στην πολύ σημαντική αρχή της μη διάκρισης ενώπιον κρατών μελών. Επομένως, ε, ε, χαιρόμαστε ιδιαίτερα για τη συζήτηση εδώ. Ελπίζουμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα μπορέσει να εγκρίνει και ένα ψήφισμα το οποίο θα αποστείλει σαφές μήνυμα για το ποιοι είναι οι στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτές τις διαπραγματεύσεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα να δώσω το λόγο στον συγητή για να ε, βγάλει τα συμπεράσματά του για τη συζήτηση. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Πάρα πολύ σύντομα. Καταρχάς να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους ε, για τις ε, παρατηρήσεις τους. Τα σημείωσα όλα και ελπίζω ότι θα συνεργαστούμε πολύ καλά όσον αφορά τις τροπολογίες. Ε, κάποιες μικρές διευκρινήσεις. Κάποια θέματα τα είχαμε θέσει ευθύς εξ αρχή ε, στην ε, έκθεση, αλλά επειδή υπήρχε ε, περιορισμός και έπρεπε να είμαστε πιο λακωνικοί, έπρεπε να κάνουμε κάποιες περικοπές και συμφωνώ μαζί σας ότι λείπουν κάποια πράγματα. Όσον αφορά τα εμπορικά θέματα, η Ευρώπη εμπορεύεται λίγο πολύ με όλο τον κόσμο και θεωρώ αδύνατο να μην έχουμε εμπορικέ σχέσει με την Τουρκία. Όσον αφορά τη θέση μου, προσωπικά δεν θα είχα κανένα πρόβλημα να εμπορεύουμε και με τη Ρωσία και να άρουμε οποιαδήποτε μορφή κυρώσεων, αλλά δεν εξαρτάται από μένα. Όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα τώρα, νομίζω ότι πρέπει να λάβουμε απάντηση από το Συμβούλιο. Ξέρω ότι ο πρόεδρος Λάγκε έστειλε επιστολή για να ε, του δοθεί μια εγγύηση, αλλά δεν απάντησαν ε, ίσως ε, θα μπορούσε να κάνει κάτι ακόμα η Επιτροπή Ίντα για να μπορέσουμε να αναβάλουμε και εμείς με την ησυχία μας ε, τη συζήτηση και την ψηφοφορία εάν μας εγγυηθεί κάτι τέτοιο το Συμβούλιο. Ευχαριστώ πολύ. Uh, this, our debate. Σας ευχαριστώ. Ολοκληρώσαμε εδώ την συζήτησή μας. και 1η Μαρτίου ε, το μεσημέρι είναι η προθεσμία για την υποβολή των τροπολογιών, λαμβάνοντα υπόψη και τον όσων είπαμε για την αναβολή όχι ε, του εν φακέλου. Ολοκληρώσαμε και το σημείο 8 τη ημερήσια διάταξη. Ε, υπό το σημείο 9 έχουμε τη συνεδρία των συντονιστών. Είναι και κλεισμένων των θυρών και θα ξεκινήσει βέβαια όπως έχει προβλεφθεί σε 35 λεπτά από τώρα, δηλαδή στις 5.30. Οπότε διάλειμμα για καφέ μέχρι τότε λοιπόν. Σας ευχαριστώ όλους για τη συμμετοχή σας.